I think we can start now, if, uh, if you could please take your seats. Let's adopt... Λοιπόν, ας υιοθετήσουμε την ημερήσια διάταξη. Όπως ξέρετε η ημερήσια διάταξη έχει ήδη σταλεί από τις προηγούμενες εβδομάδες. Θα έλεγα λοιπόν ε, να αλλάξουμε αυτή την ημερήσια διάταξη, αλλά ήθελα να σας πω ότι δεν υπάρχει το παλιό κείμενο ε, ε, και υπάρχει το καινούριο κείμενο μόνο αγγλικά και όχι στις προηγούμενες γλώσσες. Θα ήθελα όμως εδώ να προσθέσω ένα θέμα μετά το 10 το οποίο θα είναι μία ανταλλαγή απόψεων για τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2011 με εισηγητή τον κύριο Μπέρμαν. Έχετε καμία αντίρρηση ή σχόλια σχετικά με την ε, προτινόμενη τροπολογία της ημερησίας διάταξης. Αν όχι, υιοθετεί τη ημερησία διάταξη. Έχουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης 16-17 Μαρτίου, 12 Απριλίου, 10 Μαΐου. Ε, βρίσκονται μέσα στο φάκελο της συνεδρίασης. Εάν έχετε παρατηρήσεις παρακαλώ να ε, στείλετε τις παρατηρήσεις σας στη γραμματεία. Διαφορετικά θα θεωρήσουμε ότι έχουν ε, υιοθετηθεί. Έχω μόνο μία ανακοίνωση. Ορισμένοι από εσά ίσως αναρωτιούνται γιατί η ημερήσια διάταξη δεν ε, παρουσιάζει τη συνηθισμένη παρουσίαση της εισερχομένης Προεδρίας, δηλαδή της Βελγικής Προεδρίας σχετικά με τις προτεραιότητες. Θα δείτε ότι υπήρχε στο προηγούμενο κείμενο αλλά όχι στο αναθεωρημένο κείμενο της ημερήσιας διάταξης. Όταν ε, προετοιμαζόταν η Βελγική Προεδρία είχε συμφωνηθεί ότι θα ερχόταν ένας υπουργό. αλλά αυτό άλλαξε όταν ε, κατόπιν της επίσημης ε, προσκλήσεώς μας ο Υπουργός είπε ότι κατά την άποψη του Βελγίου δεν υπάρχει ρόλος στην ε, ε, εναλλασσόμενη προεδρία μετά την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Και το επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει ρόλος για την εναλλαγή της προεδρίας μετά την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας και ότι η ύπατος ε, πρόσωπος τώρα προεδρεύει το Συμβούλιο των Εξωτερικών Υποθέσεων και άρα καταρτίζει και την ημερήσια διάταξη. Και η άποψη αυτή κατά πάσα πιθανότητα ε, έχει τη σύμφωνη γνώμη της ΙΠΑ ε, του εκπροσώπου η οποία όμως δεν είναι διαθέσιμη για να μας μιλήσει σήμερα. Δεν ξέρω τι πρέπει να σας πω επί του θέματος κυρίες και κύριοι γιατί νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και ε, εάν ε, βάλετε το, ανοίξτε το κουτί της Πανδώρας ενδέχεται να δείτε ότι είναι γεμάτο σκουλίκια. Οπότε δεν ξέρω τι πρέπει να σκεφτούμε με την εναλλασσόμενη Προεδρία, τι πρέπει να σκεφτούμε ε, για το πρόγραμμα εξωτερικών υποθέσεων, αλλά ελπίζουμε ότι μέχρι τον Ιανουάριο θα έχει ξεκαθαριστεί. Εν πάση περιπτώσει, ε, η Βελγική Προεδρία είχε αποφασίσει να οργανώσει μία άτυπη συνάντηση Υπουργών Αναπτύξεως κατά τη διάρκεια του έτους και οι συντονιστές θα προτείνουν πώς θα αντιδράσει η Επιτροπή μας. Ο Επίτροπος Πίμπαλξ ε, δέχθηκε να παρουσιάσει μία ε, παρουσίαση παρόλο που ε, του το είπαμε τελευταία στιγμή αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις, την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Προεδρίας. Λοιπόν, Πρέπει ίσως να σκεφτούμε τις επιπτώσεις των σχολείων της Βελγικής Προεδρίας. Ο κύριος Γκέρενς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ανεκάλυψα ε, μάλλον ε, πληροφορήθηκα ε, όταν παρουσιάσατε το πρόβλημα του τι γίνεται. Δηλαδή υποτίθεται ότι πλέον δεν έχουμε συνομιλητή πέραν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τότε θα πρέπει να γραφεί προς την Προεδρία και να τους πούμε ότι είμαστε σε μια απαράδεκτη κατάσταση, σε μια απερίγραπτη κατάσταση όπου με τη συνθήκη της Λισαβόνας ελπίζαμε ότι θα διευκολύναμε τα πράγματα ενώ τώρα δεν έχουμε συνομιλητή. Πρέπει λοιπόν να παραπονεθούμε, να, το, να ενημερώσουμε τους πάντες και να ενημερώσουμε και την ε, ε, Προεδρία του Συμβουλίου που θα πρέπει να λάβει ένα αντίγραφο. Κατά τη γνώμη είναι απαράδεκτη η θέση αυτή. Άλλα σχόλια. Λοιπόν, συμφωνώ με αυτά που είπε ο Σάρλ. Δηλαδή, παραπέουμε. Θα ήθελα να πω γιατί το έχω πει πολλές φορές στην Επιτροπή αυτή, ότι σαν υπεύθυνο για την ανάπτυξη είχα την ίδια εντύπωση όταν ήμουν υπουργό Ανάπτυξης, διότι κατόπιν οδηγιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχαμε καταργήσει το Συμβούλιο των Υπουργών Ανάπτυξης, το οποίο ήταν απαράδεκτο. Και ο Επίτροπος ήθελε να αφήσει μόνο μία μονάδα συμβουλευτική την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε πει ότι αν δεν μπορέσουν να ακολουθήσουν όλες οι προεδρίες ε, και ε, να έχουμε τουλάχιστον μία άτυπη συζήτηση θα πρέπει να προαχθούμε κατά κάποιον τρόπο για να μπορέσουμε να έχουμε μία συζήτηση επί του θέματος. Λοιπόν, ε, πολλές εθνικές αντιπροσωπείες που ανελάμβαναν την Προεδρία, η χώρα των οποίων ανελάμβαναν την Προεδρία, οργάνωναν αυτή τη συνάντηση και πρέπει να πω ότι χαρακτηρίζω χαρακτηρίζω απαράδεκτη αυτή τη διαδικασία. Μας κοροϊδεύουν. Είναι ε, τώρα η δεύτερη φάση και νομίζω ότι είναι κάτι που το οποίο δεν μπορούμε να δεχθούμε να περάσει έτσι. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος του Συμβουλίου στην αίθουσα. Κάποιος εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Όχι. Λοιπόν, ίσως θα πρέπει να στείλουμε ένα περιστέρι με το μήνυμα στο Συμβούλιο. Συμφωνώ με τον κύριο Γκόρενς ε, και εγώ εκπλήσωμαι. Διότι είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό από το θέμα της περιστρεφόμενης προεδρίας. Είναι πολύ σημαντικό. Και όπου πάτε Παντού μας λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασκεί μαλακά την εξουσία της σε θέματα όπως η δημοκρατία κτλ. που θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Αν δείτε όμως τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, ο αναπτυξιακός προϋπολογισμός είναι αστείος Ήμασταν εκεί για να ε, προστατεύσουμε εκατομμύρια ατόμων. Δεν είναι κάποιος που κάθεται στο Στρασβούργο, ε, δουλεύουμε επί τόπου. Αλλά στο Κοινοβούλιο η εργασία η οποία κάνουμε, η πραγματική εργασία που γίνεται επί του θέματος ε, αγνοείται πλήρως. Ενώ όλες οι άλλες επιτροπές κάνουν άλλα πράγματα που δεν προασπίζονται κανέναν πουθενά ε, κανείς δεν μας παίρνει σοβαρά και μας λέγουν ότι εξασχείται μαλακά η εξουσία και υποφελείται όλος ο κόσμος, όλοι οι φίλοι από τη δουλειά μας ενώ πιστεύω ότι οι μόνες ουσιαστικές επιτροπές είναι η εμπορική, περιβαλλοντολογική και αναπτυξιακή. Εάν λοιπόν αυτές δεν μπορέσουν να επηρεάσουν την υφήλιο, θα πρέπει να μην ομφαλοσκοπούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτή την ε, εξουσία μας και οι συντονιστές να επισκεφθούν τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και να προσπαθήσουμε να ξανασυζητήσουμε μαζί του τις εξουσίες του Κοινοβουλίου και το τι πρέπει να γίνει. Οι συντονιστές θα το συζητήσουν στη συνέχεια για να δούμε ε, πώς θα ληφθεί μία απόφαση. Ανακοινώσει τη Επιτροπής. Με συγχωρείς, Σάρλ. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν θέλω να με παρανοήσετε, δηλαδή δεν τα βάζω με τη βελγική ε, αντιπροσωπεία, δεν φταίει ο Σαλ αλλά είναι η αδυναμία να εφαρμόσουν ουσιαστικά τις διατάξεις συνθήκης της Λισαβόνας. Θα πρέπει λοιπόν να διαμαρτυρηθούμε, να καλέσουμε όποιον θέλουμε και αν τον καλέσουμε ε, σαν προνομιούχο παρατηρητή της πολιτικής ε, ανάπτυξης και συνεργασίας μπορεί να έρθει να εκφραστεί. Τίποτα δεν μας ε, εμποδίζει να προχωρήσουμε με αυτό τον τρόπο. Ευχαριστώ, Τσάρλς. Όταν θα το συζητήσουμε με τους συντονιστές θα το λύσουμε και θα συμφωνήσουμε επί της πολιτικής. Ανακοινώσεις άλλες. Ε, κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να λάβει το λόγο, κάποιος από τους παρισταμένους θέλει να λάβει το λόγο, όχι. Τώρα λοιπόν έχουμε ε, μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία που είναι να προωθήσουμε τα κοινοβούλια στις αναπτυσσόμενες χώρες και να παρουσιάσουμε ε, τις ε, θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως σας είπα, ε, το Κοινοβούλιο ηγείται. Υπάρχει η μαλακή εξουσία και η σκληρή εξουσία. Προσπαθούμε όμως να βοηθήσουμε χώρες που θέλουν να προωθήσουν τη δημοκρατία στο εσωτερικό τους. Και γι' αυτό θα δώσω αμέσως το λόγο στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το γραφείο της προωθήσεως της Δημοκρατίας, τον κύριο Ντίκ Τούνστρα, που θα μας ενημερώσει για τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του γραφείου του και για το τι έχει πράξει και ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Έχετε 10 λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα Ε, διότι η Επιτροπή σας συνδέεται στενά με τις εργασίες μας. Έχουμε ήδη συνεργαστεί στενά από πέρυσι, όταν η Επιτροπή σας και οι συνάδελφοι από τη Γραμματεία της Επιτροπής συνεργάστηκαν μαζί μας για την εκπόνηση ενός ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας σε εξωτερικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία σήμερα να σας παρουσιάσω το γραφείο προώθησης της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ας μιλήσουμε για το ιστορικό υπόβαθρο. Γιατί αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συγκροτήσει μια τέτοια υπηρεσία. Ο τίτλος είναι Γραφείο Προώθησης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, OPPD, Ε, και ανταποκρίθηκε το Κοινοβούλιο σε αυξανόμενο αριθμό αιτήσεων ε, για αερογή προς τις νέες και αναδυόμενες ε, δημοκρατίες, όπως ονομάζονται. Επίσης προς ευπαθή κράτη που απέρχονται από σειράξεις, παραδείγματος χάρη, από κρίσεις και ο στόχος είναι η στήριξη των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Στην αρχή δεν ξέραμε πώς να χειριστούμε αυτόν τον αυξανόμενο αριθμό αιτήσεων και λειτουργούσαμε ad hoc, κατά περίπτωση. Το 2006 διοργανώθηκε μία διάσκεψη των Προέδρων των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων ε, στην Κοπενχάγη και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από τα 27 κράτη-μέλη κάποια εθνικά κοινοβούλια είχαν συμμετάσχει έμεσα ή άμεσα σε τέτοια προγράμματα. Στη Γερμανία, παραδείγματο χάρη, στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω του Ιδρύματο του Westminster και στην Γαλλία μέσω τη Γερουσία ε, υπήρχαν τέτοια προγράμματα κοινοβουλευτική στήριξη και άρα η διάσκεψη κατέληψε στο πόρισμα ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα υπηρεσία για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ε, αυξανόμενες αιτήσει. Η δημοκρατία φυσικά είναι πολύ ευρύτερη έννοια πέρα από τον ίδιο τον κοινοβουλευτικό θεσμό. Ε, και ε, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς το λαό αλλά και τίποτα δεν διαρκεί χωρίς ε, τα θεσμικά όργανα. Οπότε θα πρέπει εμείς να ασχοληθούμε με τον εκδημοκρατισμό και τη δημιουργία θεσμικών οργάνων σε αυτές τις νέες δημοκρατίες. Δηλαδή χρειαζόμαστε συνομιλητές σε αυτές τις χώρες. Φυσικά λαμβάνουμε πλήρως υπόψη την ανάγκη που υπάρχει να εμπλακεί άμεσα και η κοινωνία των πολιτών διότι ξαναλέω η δημοκρατία δεν περιορίζεται περιορίζεται μόνο σε μια κοινοβουλευτική συνέλευση. Χρειαζόμαστε ανθρώπινους πόρους, χρειαζόμαστε οικονομικούς πόρους, δεν μπορούμε να καλύψουμε όλες τις διαστάσεις του ζητήματος, οπότε επικεντρωθήκαμε ε, στους συνομιλητές που θα έχουμε στις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις αυτών των χωρών. Εδώ και δύο χρόνια, ε, από το 2008, έχουμε αρχίσει επιτόπου επιχειρήσεις ε, και ευδοκίμησαν οι προσπάθειές μας προς το παρόν. Ε, τώρα αναπτύσσονται αυτοί οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί και το σημαντικό διαπιστώσαμε είναι η εμπιστοσύνη. Να έχουμε σχέση πραγματικών ομοτήμων. Αυτό είναι ένα στοιχείο κλειδί της διαδικασίας και δείχνει ιδιαίτερη προθυμία οι ομοτήμοι μας να συνεργαστούν μαζί μας. Δεν έχουμε τακτικούς ε, δωρητές, ε, δεν έχουμε ε, συμβάσεις αν θέλετε, δεν αγοράζουμε κάτι, δεν είναι αυτό ο στόχο μα. Ε, θέλουμε να υποστηρίξουμε τι ενδογενεί ικανότητε αυτών των χωρών ε, και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε μακρόπνη συνεργασία με αυτέ τι ε, κοινοβουλευτικέ συνελεύσει ενδιαφέρονται οι ομότιμοι μας ε, να αντλήσουν διδάγματα από την εμπειρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ και 50 ε, χρόνια ε, που από μια κοινοβουλευτική συνέλευση μεταξελίχθηκε σε σύνομο θέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2007 λοιπόν συγκροτήθηκε αυτή η νέα υπηρεσία και τώρα έχουμε αποκτήσει ήδη κάποια εμπειρία από τις επιτόπου επιχειρήσεις μας έχουμε καταλήξει σε κάποιο είδους ε, ε, μεθοδολογία δράσης. Το κοινοβούλιο, τα κοινοβούλια πρέπει να ζητήσουν αρρωγή. Σε αυτό έγινε η μεθοδολογία μας. Ε, δεν πηγαίνουμε εμείς ανά τον κόσμο και του ρωτάμε, χρειάζεστε βοήθεια, χρειάζεστε υποστήριξη. Εκείνοι στρέφονται προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμείς δείχνουμε προθυμία να τα επικουρήσουμε. Τα ίδια τα κοινοβούλια λοιπόν πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματά τους. Εμείς παρεμβαίνουμε μόνο όταν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει σοβαρή δέσμευση εκ μέρους τους να μεταμορφώσουν την κοινωνία τους σε μια εκδημοκρατισμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Μαζί με τους λοιπούς δωρητές ε, προσπαθούμε να κάνουμε μία μοναδική αξιολόγηση σχετικά με την ε, βοήθεια που μπορεί να προσφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πλήρη διαφάνεια και σε ανοιχτή συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους δωρητές που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη χώρα. Φυσικά συνεργαζόμαστε με τους ε, συναδέλφους από τις αντιπροσωπείες Ευρωπαϊκής Ένωσης αν υπάρχουν στη συγκεκριμένη χώρα για να έχουμε μια κοινή προσέγγιση και δεν αποσκοπούμε στην κάλυψη όλων των διαστάσεων που προβάλλει το, ε, το εκάστοτε κοινοβούλιο ως ανάγκη του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν δύναται ε, να παράσχει τέτοιου είδους ε, σφαιρική βοήθεια. Προσπαθούμε λοιπόν μετά την αξιολόγηση να χορηγήσουμε κονδύλια και να υποστηρίξουμε προγράμματα ε, από αυτούς που είναι σε καλύτερη θέση για να υποστηρίξουν το στόχο μας. Επίσης έχουμε τακτικές ε, συνεδριάσεις ε, συντονισμού της δράσης των δωρητών για να γνωρίζουμε τι θα γίνει στο συγκεκριμένο κοινοβούλιο. Και το εκάστοτε κοινοβούλιο φυσικά ε, θα πρέπει να έχει μια ε, διαφανή στάση και να μην προσπαθεί να στρέψει τον έναν δωρητή κατά του άλλου ε, για να αποκομίσει τα μέγιστα ωφέλη. Επίσης, χρησιμοποιούμε μέτρα σύγκρισης. Μπορεί να μην ακούγεται και τόσο σημαντικό. Αλλά ξέρετε για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε τέτοια κοινοβούλια ε, εισερχόμεθα σε μια σχετικά καινοτόμη διαδικασία. Υπάρχουν πολλοί δωρητές, πολλοί οργανισμοί που κρίνουν πως ε, ε, χρειάζεται έρευνα σχετικά με την εκπόνηση μέτρων σύγκρισης για την αρρωγή προς το Κοινοβούλιο, για να κάνουν και αυτοαξιολογήσει στα Κοινοβούλια. Προσπαθούμε να τους ε, δίνουμε πρότυπα που μπορούν να χρησιμοποιούν τα ίδια τα Κοινοβούλια για να αναλύσουν την κατάστασή τους σε σχέση με το ε, συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο ε, που έχουν εκπονήσει. και προσπαθούμε να προσφέρουμε και κάποια πολιτική καθοδήγηση στα πλαίσια αυτού του συνολικού αναπτυξιακού σχεδίου. Um, we have, Η υπηρεσία μας έχει ένα πρόγραμμα δράσης που βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες, ας το πούμε έτσι. Πρώτον, ε, η υποστήριξη τεχνικού χαρακτήρα, η τεχνική αρρωγή δηλαδή. Σας ε, είπα ότι προσπαθούμε να κάνουμε και κάποια έρευνα, ε, να έχουμε δημοσιεύσεις. Ταυτόχρονα όμως εξακολουθούμε να ασκούμε πίεση σε, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ίδιο στόχο, έτσι, για την υποστήριξη της δημοκρατίας, για να παραμένει ύψιστη προτεραιότητα στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα καλό παράδειγμα είναι ότι σε συνεργασία με τη δική σας Επιτροπή, την Υποεπιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, έχουμε δραστηριοποιηθεί και έχουμε παίξει καταλητικό ρόλο για την δημιουργία των συμπερασμάτων του Συμβουλίου που εγκρίθηκαν τον Οκτώβρη πέρσι ε, μετά το ε, σχετικό, το αντίστοιχο ψήφισμα μάλλον του Κοινοβουλίου που επίσης εκπονήθηκε πέρσι τον Οκτώβριο. Κατόπιν, προσπαθούμε να ε, με μια ε, συνεργασία μάλλον θεσμικού χαρακτήρα με άλλους δωρητές όπως το Ίδρυμα ε, Westminster, το Γερμανικό Stiftung, ε, το UNDP, του ΟΗΕ και με όλους τους υπόλοιπους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς που εμπλέκονται στις δραστηριότητες στήριξης κοινοβουλευτικής δραστηριότητας. Το πιο σημαντικό που έχουμε κάνει είναι μια στρογγυλή τράπεζα ε, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι από διάφορα think tanks ε, δεξαμενές σκέψεις, συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάποιοι βουλευτές ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόσο ώστε να υπάρξει ένας προβληματισμός σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας ε, των κοινοβουλευτικών συνελεύσεων, δηλαδή έγιναν συζητήσεις σχετικά με, το με τη συγκεκριμένη παρακολούθηση που ήδη προβλέπεται ή θα πρέπει να προβληθεί για να δοθεί συνέχεια στα συμπεράσματα του Συμβουλίου που εγκρίθηκαν πέρυσι τον Οκτώβριο. Γιατί ουσιαστικά δεν έχουν γίνει και πολλά πράγματα από πέρυσι τον Οκτώβριο για διάφορους λόγους ε, καθυστερήσεις σε σχέση με την έγκριση της ε, συνθήκης της Λισαβόνας. Ε, όλοι επικεντρώθηκαν ε, στη συνθήκη της Λισαβόνας ή ασχολήθηκαν μόνο με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων η ουσία είναι ότι δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα, δεν έχει δοθεί ουσιαστική συνέχεια στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και αυτό πρέπει να γίνει γιατί όπως γνωρίζετε ε, ε, μία νέα συνεδρίαση του Συμβουλίου για τη συνέχεια για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου έχει προβλεφθεί ήδη για τον Νοέμβριο του 2010. Από την εμπειρία μας ε, δε κρίνουμε πως υπάρχει μία δυναμική ούτως ώστε, όπω σα έλεγα, να είναι μεγάλη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση η στήριξη κοινοβουλευτική ε, δραστηριότητας ε, και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια αντίστοιχη προθυμία από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υποστήριξη αυτή τη διαδικασία. Αυτό λοιπόν είναι, αυτά είναι τα βασικά στοιχεία στο ψήφισμα του ΕΛΚ όπως ψηφίστηκε τον Οκτώβριο και Στη συνέχεια είχαμε τη συμπεράσματα του Συμβουλίου τον Νοεμβρίου. Υπάρχει μια σειρά δραστηριοτήτων όπου εμείς ως γραφείο προσπαθούμε να βοηθήσουμε και την Επιτροπή ε, Ανάπτυξης ως προς την χρηματοδότηση και στα κοινοβούλια των νέων αναδιωμένων δημοκρατιών, ιδιαίτερα από την Αφρική. Και θεωρούμε ότι στη μεγάλη πλειοψηφία στη πλειοψηφία τους αυτές οι χώρες δεν ήξεραν ότι υπάρχει χρηματοδοτική υποστήριξη. Αν λοιπόν θέλουμε να παραμείνουμε αξιόπιστοι σε αυτό το τομέα, τότε καθίσταται σαφές ότι τα κράτη ε, που μπορούν να τύχουν χρηματοδοτικής υποστήριξης θα πρέπει να ενημερωθούν έτσι ώστε να ασκήσουν το δικαίωμά τους εποπτείας ως προς το εκτελεστικό σκέλος. Επίσης ως προς το δημοκρατικό έλεγχο στα περιφερειακά έγγραφα στρατηγικής και σε αυτό το τομέα θα θέλαμε να συνεργαστούμε με τη γραμματεία της Επιτροπής και τέλος οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής συνεργασίας είναι ένας άλλος ε, βασικός τομέας, έτσι ώστε να προβούμε προς ε, τεχνική αρρωγή, έτσι ώστε οι συνάδελφοι που εργάζονται στα κοινοβούλια να καταρτίζονται, έτσι ώστε να μπορέσουν να μπορέσουν να διαπραγματευτούν αυτό το πλαίσιο συμφωνιών. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα φτάσουμε σε, κάποιο, κάποια συμπεράσματα στο δεύτερο ημισή του έτους. Μετά το ψήφισμα του Οκτωβρίου και πριν από αυτό, φτάσαμε σε ένα συλλογικό επίπεδο συνεργασίας με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσης θα προβάλλουμε κατάρτιση στους συναδέλφους της ε, κοινοτικής αντιπροσωπείας, διότι όσο και να σας εκπλήσει, σε πολλές κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες δεν υπάρχουν εμπειρογνώμονες που να μπορούν να καλύψουν θέματα σχετιζόμενα με τη δημοκρατία. Δεν ε, δίνεται αναφορά ως προς την κατάσταση πραγμάτων, ως προς τη δημοκρατική εξέλιξη αυτών των χωρών και ε, οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν το, θεωρήσουν, δεν το θεωρούν ε, θέμα άμεσης προτεραιότητας. Πολλές φορές για πολιτικούς λόγους. Όμως, σε πολλές αντιπροσωπείες, όμως πολλές αντιπροσωπείες δεν έχουν επαρκές προσωπικό έτσι ώστε να το λάβουν υπόψη. Εάν εμείς θέλουμε να παραμείνουμε αξιόπιστοι ως προς τους εταίρους μας και αν ε, μιλάμε για τις ιδρυτικές αξίες, θεμελιώδεις αξίες και αν υπάρχουν ε, άρθρα της συνθήκης που μας ε, επιβάλλουν να λάβουμε υπόψη αυτές τις αξίες στην ΚΕΠΑ, νομίζω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε επαρκές προσωπικό στις αντιπροσωπείες που να καλύπτουν αυτούς τους τομείς και να μας ε, ε, μιλάνε για τα αποτελέσματα. Το ίδιο αφορά και τη χρηματοδότηση, τη χρηματοδότηση των αποστολών παρατηρητών για τις εκλογές. Πολλές φορές υπάρχουν λεπτομερείς εκθέσεις με μια πλήρη σειρά συστάσεων, αλλά μόλις εγκριθούν ε, μπαίνουν σε ένα ντουλάπι τις βάζουμε στο σιρτάρι, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Πολλοί που προεδρεύουν αυτών των ε, αποστολών παρατηρητών για τις εκλογές παραπονούνται ότι δεν συμβαίνει τίποτα με αυτές τις ε, εκθέσεις και θα θέλαμε οι ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες να λάβουν, να λάβουν πιο σοβαρά υπόψη αυτές τις συστάσεις. Τέλος, υπάρχει άλλη μια διαφάνεια. Η τελευταία. Έχουμε ορισμένα προβλήματα τεχνικής φύσης. Η τελευταία παρατήρηση αφορά το τι ε, αποκομίζουμε, το τι ε, παραδίδουμε, ποιο είναι το έργο μας. Δηλαδή, τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο έργο για την ευμερία των πολιτών, τότε δεν μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για ένα βιώσιμο σχέδιο. Άρα αυτό που κάνετε εσείς είναι ύψης της ε, σημασίας για την ε, μεγαλύτερη ε, αξιοπιστία της πρόθεσης της δημοκρατίας. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρούμε μια καλύτερη εξισορρόπηση ως προς το ρυθμιστικό πλαίσιο, τις ρυθμιστικές αξίες και την Realpolitik. Πολύ συχνά κινούμαστε εντάχει προς την Realpolitik και κλείνουμε τα μάτια μας ως προς τις αξίες που είναι εγγεγραμμένες και στην συνθήκη. Άρα, για να ε, προωθήσουμε αυτό το θέμα του πυρήνα της δημοκρατίας, είναι ύψης της σημασίας Πιστεύω ότι αυτό είναι ε, η πεμπτουσία των στόχων μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τούνστρα. Η Φραντσέσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Έχω αρκετές ερωτήσεις. Ε, την πρώτη ερώτηση, πρώτη ερώτηση, κάτι που ίσως δεν άκουσα καλά, ως προς θέμα της ε, δημοσιονομικής υποστήριξης δεν ξέρω κατά πόσο ενισχύουν τα κοινοβούλια ή όχι. Το συζητήσαμε και αλλού. Πώς το αποτιμάτε, πώς το αξιολογείτε. Επίσης είπατε ότι η δημοκρατική υποστήριξη θα πρέπει να αναφέρεται πολύ περισσότερο στα ε, έγγραφα στρατηγικής για τις χώρες. Όταν εφαρμόζουμε αυτά τα έγγραφα στρατηγικής, τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε. Έμπρακτα επιτοπίως δηλαδή για να ενισχύσουμε τις δημοκρατίες, ιδιαίτερα το ρόλο του κοινοβουλευτισμού και πώς βλέπετε την, ε, το, τη Διακυβουλευτική Επιτροπή Ίσης Εκπροσώπησης. Στα τελευταία σας λόγια είπατε ότι θα πρέπει να είμαστε συνεπείς στις πολιτικές μας. Ποια είναι τα ε, πιο χτυπητά παραδείγματα που υποσκάπτουν τον κοινοβουλευτικό δημοκρατικό ρόλο. Πολύ καλές ερωτήσεις, Φραντσέσκα. Κάποιος άλλος, έχω και εγώ μία ερώτηση, αλλά θα περιμένω να ακούσω πρώτα τους άλλους συνοδέλφους. Μετά την ερώτηση του κ. Κέλλαν, μπορώ να πω ότι υπάρχει ένα ευεργέτημα ε, εάν αυτός ο οργανισμός, αυτό το γραφείο μπορεί να ενισχύσει τον ρόλο άλλων κοινοβουλίων ως προς τις επιτροπές ε, λογοδοσίας, διότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε ως προς την ε, δημοσιονομική υποστήριξη είναι ότι πολλές φορές πολλά από τα χρήματα ε, που χορηγούμε δεν ξέρουμε κατά πόσο τα πανήθηκαν όπως ε, θα θέλαμε επειδή δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτή τη διαδικασία. Οι βουλευτές στην εν λόγω χώρα θα πρέπει να έχουν ένα μηχανισμό λογοδοσίας. Αν υπάρχουν, αν γίνεται κάποια χειραγώγηση και να ζητήσουν ας πούμε κάποια λογοδοσία για, το, για τα έξι ή πέντε νοσοκομεία που έπρεπε να χτιστούν και δεν χτίστηκαν. Να υπάρχει μια επιτροπή λογοδοσίας δηλαδή. Και ίσως θα εξοικονομήσουμε πολλά χρήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευεργέτημα θα ήταν πολύ μεγάλο γιατί θα μπορούσαν να μας πούν ότι είναι ευτυχής ή όχι με αυτή τη διαδικασία. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να ενισχυθούν αυτές οι πτυχές σε αυτά τα κοινοβούλια, δηλαδή να υπάρχει μια επιτροπή λογοδοσίας και επιτροπές ελέγχου των λογιστικών βιβλίων για να δουν πώς δαπανούνται, πώς δαπανούνται αυτά τα κονδύλια και αν δαπανούνται σωστά. Ευχαριστώ. Σε σχέση λοιπόν με την υποστήριξη της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, ε, ήθελα να ρωτήσω αν έχετε σκεφτεί με ποιο τρόπο μπορούν τα αφρικανικά ε, κοινοβούλια να συμμετάσχουν στον ευρύτερο κοινοβουλευτικό διάλογο. Σήμερα συζητήσαμε με το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και την Κοινωνία των Πολιτών κατόπιν πρωτοβουλία της Επιτροπής και συζητήσαμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να πλουστεύσουμε αυτή τη διαδικασία διαλόγου και συζητήσαμε όλο ιδιαίτερος ε, το ρόλο των ε, κοινοβουλίων. Αυτό ήταν ενδιαφέρον για τα κοινοβούλια, γιατί θα όσοι προέρχονται από ε, δημοκρατίες που δυσλειτουργούν θα μπορούσαν να συναντηθούν με βουλευτές δημοκρατιών που λειτουργούν εύρυθμα. Και Επίσης, ε, στα πλαίσια των περιφερειακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε σχέση με τις ε, συμφωνίες ε, οικονομικής εταιρικής σχέσης, θα μπορούσαμε να επιτύχουμε μια στενότερη συνεργασία ανάμεσα στα κοινοβούλια. Αυτό θα μας ενδιέφερε και μας. Δηλαδή, στα πλαίσια μιας εταιρικής σχέσης θα μπορούσαμε να δούμε, να διαπιστώσουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να διευρύνουμε τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης ε, στα κοινοβούλια των Αφρικανικών χωρών. Λοιπόν, καταρχήν ε, ευχαριστώ κύριε Τόνστρα για την έκθεσή σας και πιστεύω ότι είναι μια έκθεση η οποία διευκρινίζει πώς ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να επιτύχει τους ε, στόχους της για την πρόθεση της ε, δημοκρατίας και της ορθής διακυβέρνησης και πώς μπορεί να τα εφαρμόσει στην πρακτική. Αυτό που είναι βασικό για μας στην Επιτροπή, όπως άλλωστε και στις αντιπροσωπείες και στην παρακολούθηση των εκλογών, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να φροντίσουμε οι αντιπροσωπείες να έχουν ε, συγκεκριμένες εντολές να παρακολουθούν ε, την ε, εξέλιξη της δημοκρατίας και την εργασία της κυβέρνησης και όταν καταρτίζεται μία έκθεση για το Κοινοβούλιο να μπορεί το Κοινοβούλιο στη συνέχεια να την επεξεργάζεται. Δεν μπορεί το Κοινοβούλιο να λειτουργήσει μόνο του. Πρέπει να υπάρχει μια εξελικτική διαδικασία και γι' αυτό ή στο μέλλον όταν υπάρχουν ταξίδια αντιπροσωπιών ή παρακολούθηση εκλογών θα πρέπει να προσέξουμε συγκεκριμένα και να επιτηρήσουμε τις εξελίξεις και να επαληθεύουμε σε τακτά διαστήματα τα θέματα αυτά. Επίσης αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να υπάρχει υπάρξει ένα είδος benchmarking, βαθμολογήσεως, δηλαδή να αξιολογούμε πώς αναπτύσσεται η δημοκρατία, πώς εφαρμόζονται οι κοινοβουλευτικοί κανόνες και θα ήθελα να ξέρω τι ε, όργανα έχουν προβλεφθεί για τη βαθμολόγηση αυτή, για το benchmarking, για να μπορέσει κανείς να αποκομίσει και τα δέοντα συμπεράσματα. Προτού να απαντήσει ο Ντίκ, ε, θα ήθελα να εμπλέξω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πω και κάτι προς τους συναδέλφους. Ο κύριος Τρούντσα είπε ότι πολλές φορές δεν είμαστε συνεκτικοί και ξεχνούμε τη δημοκρατία. Διότι η ομόλογος χώρα με την οποία συζητούμε έχει διαφορετικό σύστημα και πλέον δεν συζητάμε για δημοκρατία, όπως παραδείγματο χάρη στην Κίνα. Η Κίνα είναι ένας ουσιαστικός νέος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τελευταίος ε, δημοσιεύθηκε ένα βιβλίο κινέζικα για το πώς λειτουργούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, πώς εκλέγονται οι ευρωβουλευτές, πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι επιτροπές, πώς οι βουλευτές καταλήγουν στα ψηφίσματα και τι συμβασμούς κάνουν και το, γραφείο, το βιβλίο αυτό λοιπόν έχει ε, γραφεί αυτή κινέζικα θα διδάσκεται στα πανεπιστήμια και θα διαβάσουν πώς εμείς ε, ε, κάνουμε τις δουλειές μας εδώ, πώς εκλεγόμαστε κτλ. Και οι Κινέζοι είναι πολύ ικανοποιημένοι και επέτρεψαν να εκδοθεί το βιβλίο αυτό. Δηλαδή ε, ε, υπάρχει μια ε, αποστολή η οποία είναι ευαίσθητη αλλά εγώ θα πάω την επόμενη εβδομάδα στο Πεκίνο για την έκδοση επισήμως αυτού του βιβλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοί μου θέλουν κάτι να πούνε. Εγώ ήθελα απλώς να απαντήσω εν συντομία σε δύο-τρία σημεία και ίσως θα ξεκινήσω λέγοντας ότι είχα την τιμή να βοηθήσω με το πρόγραμμα για την αντιπροσωπεία της ΕΚΟΒΑΣ προσφάτως και πρέπει να σας πω ότι ε, σαν εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος απευθύνεται εις ε, βουλευτές ε, Αφρικανούς βρήκα ότι ήταν πολύ χρήσιμο. Δεύτερον, το θέμα των αντιπροσωπιών και των ταξιδιών που αναφέρθηκε. Προφανώς έχουμε την διακυβέρνηση σαν ουσιαστικό θέμα σε όλα τα θέματα συνεργασίας μας είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ και οι αντιπροσωπείες εξετάζουν το θέμα αυτό καθημερινά και πρέπει να τονίσουμε και να πούμε ότι οι αντιπροσωπείες αν ε, δεν έχουν ε, αρκετές δυνατότητες ε, δεν πρέπει να προεξοφλούμε ότι δεν χρησιμοποιούμε και δεν εφαρμόζουμε τη σωστή διακυβέρνηση. Αντιθέτως προσπαθούμε να εντάξουμε το εθνικό σύστημα ελέγχου και το επαναλαμβάνω και δεν αναφέρουμε μόνο στη δυνατότητα του Εθνικού Κοινοβουλίου Κοινοβουλίου να ελέγχει τις δημόσιες δαπάνες αλλά επίσης και την ανώτατη ελεγκτική αρχή και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τα μέσα ενημέρωσης που είναι θέματα που παρακολουθούμε, μας ανησυχούν και είναι ένα βασικό στοιχείο της πολιτικής μας. Πρέπει να σας πω ότι τα θέματα αυτά έχουν συζητηθεί επανειλημμένως με την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πολύ συχνά τους προμηθεύουμε πληροφορίες σχετικά με τα πορίσματά μας. Δεν ξέρω αν οι συναδελφοί μου θέλουν κάτι να προσθέσουν. Ευχαριστώ. Είμαι από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ EuroPaid. Θα θέλαμε να σας δώσουμε κάποια νέα στοιχεία σχετικά με το προσωπικό συγκεκριμένα στη διαδικασία κοινοβουλευτική στήριξη. Υπάρχει ένα εγχειρίδιο που ολοκληρώνεται τώρα για το προσωπικό των αντιπροσωπιών και τα επιτόπου γραφεία. Είναι ένα ε, εργαλείο μεθοδολογικού χαρακτήρα για την διεξαγωγή επιχειρήσεων ε, στις δράσεις στήριξης ε, Επίσης έχουμε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο πάλι για το προσωπικό των αντιπροσωπιών και των επιτόπου γραφείων. Συνεργαζόμαστε δε με το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα με την υπηρεσία OPPD για την πρόθεση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και θα ενισχύσουμε τη συνεργασία με το OPPD ε, κυρίως ως προς την αξιολόγηση των αναγκών ή για τη στρατηγική καθοδήγηση και την τεχνική πραγματογνωμοσύνη ε, που, των συναδέλφων που δραστηριοποιούνται επί τόπου. Ευχαριστώ, λέει Υπάρχει κάποιο άλλος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Όχι. Ας ακούσουμε λοιπόν τις απαντήσεις ε, τώρα του κυρίου Τούστρα. Ε, για την ε, δημοσιοοικονομική στήριξη Όταν ε, λαμβάνουμε ένα αίτημα από ένα κοινοβούλιο για γενική στήριξη, εμείς εστιάζουμε στην, στον έλεγχο, στο δημοσιονομικό έλεγχο. Γιατί δείτε την ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα αυτό δεν ενεπλάκει εξ αρχής στην ομοθετική διαδικασία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά εξ αρχής ενίσχυσε την ικανότητά του ε, να παρακολουθεί τα προγράμματα, να παρακολουθεί τον προϋπολογισμό που εκτελούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε, ο έλεγχος του προϋπολογισμού πρέπει να ενισχυθεί, γιατί έτσι ενισχύεται συνολικότερα ο ρόλος του κάθε κοινοβουλίου. Αυτό είναι προτεραιότητα για μας. Συνεργαζόμαστε στενά με την ε, Παγκόσμια Τράπεζα που έχει ένα ειδικό πρόγραμμα για την ε, υποστήριξη αυτής της διάστασης κοινοβουλευτικής ζωής, ε, δηλαδή του ελέγχου. συνεργαζόμαστε στενά με την UNDP, τον απτυξιακό πρόγραμμα του ΟΗΕ, για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Επίσης προσφέρουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια στο προσωπικό για ε, το θέμα αυτό. Έτσι, ε, συμβάλλουμε στην αλλαγή των εσωτερικών κανονισμών των κοινοβουλίων, ούτως ώστε, και τώρα σας μιλάω για τα εθνικά κοινοβούλια, ούτως ώστε λοιπόν μέλη της αντιπολίτευσης ε, να, είναι, να προεδρεύουν στην Επιτροπή των Δημοσίων Λογαριασμών ή όπως ονομάζεται σε κάθε κοινοβούλιο, διότι έτσι ενισχύουμε την ε, θεσμική σημασία των εκθέσεων που προέρχονται από αυτήν την ε, Επιτροπή και τονώνεται και ο θεσμικός ρόλος ε, του Κοινοβουλίου ως προς την εποπτεία, ως προς τον έλεγχο και θεωρούμε ότι είναι ένας από τους βασικούς ρόλους κάθε Κοινοβουλίου ο έλεγχος. Αυτά για τις συνέπειες της άμεσης στήριξης. Βέβαια, ε, δεν έχουμε πάντοτε αξιόπιστες ε, πληροφορίες από πλευράς ε, των κοινοβουλίων, δηλαδή σε τι χρησιμοποιήθηκε η χρηματοδοτική στήριξη. Θέλουμε να ενισχύσουμε τον έλεγχο, αλλά ξέρετε συχνά τα εθνικά κοινοβούλια δεν έχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες, δεν ξέρουν τι πρέπει να ελέγξουν με λίγα λόγια. Έγραφα στρατηγική τώρα. Υπάρχει πάντοτε μέσα σε αυτά ρήτρα εκδημοκρατισμού πέρα από την εξακρίβωση των εκθέσεων που παίρνουμε από τα think tanks, από τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, από μη κυβερνητικές οργανώσεις, αυτό που θα επιθυμούσαμε εμείς είναι οι αντιπροσωπείες επί τόπου να ε, θεωρήσουν ε, ότι ε, είναι ιδιαίτερα σοβαρές αυτές οι ρήτρες εκδημοκρατισμού που υπάρχουν μέσα στα έγγραφα στρατηγικής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι ένας από τους αποδέκτες, δηλαδή να ενημερώνεται το Κοινοβούλιο ε, τακτικά για την κατάσταση ως προς τη δημοκρατία σε κάθε χώρα που στηρίζουμε. Ταυτόχρονα θα θέλουμε, να θέλουμε να προωθήσουμε τις διακοινοβουλευτικές επιτροπές, ε, σε... είτε μιλάμε για, περιφε... σε... για διακοινοβουλευτικές ε, ε, συνελεύσεις σε περιφερειακό επίπεδο, είτε όχι. Συνεργαζόμαστε με, τις... με την ΕΚΟΒΑΣ, όπως σας είπαμε, με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, με, τις... με την Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών, Και γι' αυτό, α και ξέχασα να σας μιλήσω και για τη Λατινική Αμερική. Οπότε τρεις ή τέσσερις φορές ετησίως ε, λαμβάνουμε ενημέρωση από αυτές τις περιφερειακές ομάδες ε, και οι ίδιες πληροφορίες θα πρέπει να υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτω ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε πώς λειτουργούν τα επιτόπου προγράμματα από θεσμικής πλευράς και για να μπορέσουμε τελικά να αναπτύξουμε τις ενδογενείς ικανότητες ε, αυτών των κοινοβουλίων. Μιλήσατε επίσης ε, για τη συνοχή των δράσεων. στα ίδια τα συμπεράσματα του Συμβουλίου αναφέρεται ότι δεν υπάρχει αγαστή συνεργασία ανάμεσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τη. Συμβαίνει αυτό και μάλιστα συμβαίνει τακτικά. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις αντιπροσωπείες της ή ένας επίτροπες. παραδείγματος χάρη, διαπραγματεύεται με μια χώρα ταυτόχρονα δε ε, διεξάγονται διαπραγματεύσεις από πλευράς ενός κράτους μέλους. Το πιο χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα είναι ε, η συνεργασία που σας είπα, που προσπαθούμε να εγκαθιδρύσουμε με κάθε χώρα, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν άλλοι δωρητές ή άλλα κρατημένα που προσπαθούν να πουλήσουν σε εισαγωγικά το δικό τους πρότυπο, το δικό τους μοντέλο. Αυτό δυσχεραίνει φυσικά ε, τη δράση μας. Και αυτό έχει αναγνωριστεί από το Συμβούλιο των Υπουργών και αναφέρεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Ένα από τα συμπεράσματα ήταν ακριβώς αυτό, ότι χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια ε, στις δραστηριότητες που έχουν αφενός η Ευρωπαϊκή Ένωση για φετέρου στα κράτη-μέλη της Ένωσης και πρέπει να υπάρχει συνεργασία και επιτόπου ανάμεσα στους δύο. Τα Αφρικανικά Κοινοβούλια, νομίζω ότι ήδη απάντησα στον Σάρλ Γκέρενς προσπαθούμε ε, να ε, ακολουθούμε τα ε, αιτήματά τους. Το γραφείο του GPA έχει ήδη δεχτεί το αίτημα των Αφρικανικών Κοινοβουλίων και προσπαθούμε να δώσουμε συγκεκριμένη συνέχεια στο αίτημά τους. Η υπηρεσία μας συμβάλλει επίσης στην εκπόνηση εγγράφων ε, για τα, τους βουλευτές που συμμετέχουν στις αντιπροσωπείες ή που συμμετέχουν σε αποστολές παρατηρητών για τις εκλογές. Κατόπιν γίνεται debriefing, ενημέρωση και ε, διαπιστώνουμε ποια είναι τα συγκεκριμένα στοιχεία της παρέμβασής μας. Τώρα για το benchmarking, τα μέτρα σύγκρισης. Στην πράξη τι κάνουμε. Κάνουμε μία καταγραφή των αναγκών του Κοινοβουλίου για να μπορέσει να λειτουργήσει εύρυθμα και κατόπιν μετά από αυτήν την τεχνικού χαρακτήρα απογραφή καταλήγουμε σε μέτρα σύγκριση, ούτως ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο να μπορεί να κάνει την αξιολόγηση σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα και τι πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης των τεχνικών ικανοτήτων του Κοινοβουλίου. Έτσι είναι ευκολότερο για μας εμάς. Όταν λέω εμάς εννοώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους συναδέλφους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τους συναδέλφους από το Ίδρυμα του Westminster ή την ε, Σουηδική, ε, τον Σουηδικό Οργανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας ή το Γερμανικό Stiftung. Έτσι λοιπόν εμείς, όλοι εμείς, μπορούμε να συμβάλλουμε και να καταλήξουμε στο πρόγραμμα που ενδείκνεται για κάθε χώρα, για κάθε συγκεκριμένο κοινοβούλιο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας αυτή, αυτή η χρήση των μέτρων σύγκρισης. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ε, μία ιστοσελίδα, μία διαδικτυακή πύλη στα πλαίσια του Κοινοβουλίου. Δηλαδή ας πούμε ότι πάω στη Μπουρκίνα Φάσο για να δω την διάρθρωση του Κοινοβουλίου και υπάρχει ένα checklist. Θέλουμε να ξέρουμε κατά πόσο υπάρχει μηχανογράφηση. Υπάρχουν στοιχεία των βουλευτών στο διαδίκτυο. Υπάρχει διαδικασία εποπτείας. Υπάρχει δηλαδή ένας απογραφικός ε, ε, κατάλογος ελέγχου. Απάντηση. Όπως σας είπα και νωρίτερα, υπάρχει περιορισμένο εύρος. Αυτή τη στιγμή διευρύνουμε το δίκτυο intranet, αλλά συνεργαζόμαστε με μια σειρά οργανώσεων και πρόσφατα έχουμε αναπτύξει μια διαδικτυακή πύλη αγορά Άγκορα ονομάζεται και ελπίζουμε να διαθέσουμε όλα τα συναφή στοιχεία για την κοινοβουλευτική ανάπτυξη. Υπάρχουν πολλά έγγραφα ενημέρωσης στη διαδικτυακή πύλη Αγκορά για αυτούς που εργάζονται και αυτούς που ε, υποστηρίζουν χρηματικά αυτό το σχέδιο το οποίο ξεκίνησε το Μάρτιο στο Παρίσι και ήταν ένα από τα απότοκα στοιχεία αυτής της συνάντησης. Πρόεδρος, τώρα θα πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το 6, το 7 μάλλον, μάλλον το 8, διορθώνει ο Πρόεδρος για πολλοστή φορά. Το 7 η αλλιευτική εταιρική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των νησιών του Σολομόντα. Εγώ είμαι η Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας μιλήσω για όλα αυτά τα στοιχεία. Σήμερα θα συζητήσουμε για τη συμφωνία με τα νησιά του Σολομόντα θα είμαι ιδιαίτερα ομός. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μείζον στοιχείο εκμετάλλευσης και απεικιοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως προς τις διαδικασίες, θα ήθελα να σας πω ότι είναι πολύ απογοητευτικό το γεγονός ότι η διαδικασία συνένεσης ε, πριν μάλλον από τη συνθήκη της Λισαβόνας υπήρχε συμβουλευτικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τώρα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνενέσει πριν από τη σύναψη μιας αλληλευτικής συμφωνίας. Άρα, de facto, θα πρέπει εμείς να ενισχύσουμε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο μιας συμφωνίας η οποία προσωρινά εφαρμόζεται. Αλλά είμαι της γνώμης και αν δείτε την έκθεσή μου θα συμφωνήσετε ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα πρέπει να αφορά μια διαδικασία πιστοποίησης, αλλά θα πρέπει να αντιταχθούμε σε ενδεχόμενες αποβάσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής και να κινηθούμε υπέρ του φορολογούμενου, των συμφερόντων των φορολογουμένων. Στις τελευταίες συζητήσεις που είχαμε, Γνωρίζουμε ότι στα νησιά του Σολομώντα εμείς πληρώνουμε 50 ευρώ ανά χιλιόγραμμο τόνου. Αυτός ο... 50 ευρώ ανά τόνο. Με συγχωρείτε, έκανα λάθος, λέει ο μιλητής. 65 ευρώ ανά τόνο. Ένα όμως χιλιόγραμμο πωλείται προς εμάς ο ίδιος ο τόνος σε τιμή 35 ευρώ. Άρα ένας τόνος αγοράζεται στη τιμή των 65 ευρώ και ένα κιλό πωλείται για 30 προς 30 ευρώ. Δηλαδή 100 χιλιόγραμμα πωλούν αγοράζονται ε, προς 65 ευρώ. Άρα κάποιος ε, κάνει, έχει ένα πολύ μεγάλο κέρδος κατά του φορολογουμένου με την αγορά του τόνου. Και τα νησιά του Σολομώντα δεν λαμβάνουν τίποτα από την όλη αυτή διαδικασία. Και ο τοπικός αλιές δεν λαμβάνει τίποτα και μιλάμε για ανάπτυξη μετά. με απασχολεί αυτό το ζήτημα, θα πρέπει να το διευθετήσουμε θέμα γιατί είναι σκανδαλώδες. Ως προς την ε, συμφωνία καθεαυτή μπορούμε να συνενέσουμε εάν ε, δεχτεί, δεχτούν και οι νήσοι του Σολομώντα αυτή την προσθήκη, την προσθήκη όρων διαφάνεια της διαδικασίας για να αναγνωρίσουμε το σύνολο των αλλιευμάτων. Θα πρέπει να βελτιωθεί αυτό το πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ποια είναι τα αλλιεύματα. Τα νησιά του Σολομώντα δεν ξέρουν σε, πόσο, ε, σε τι ποσό μάλλον ανέρχονται αυτά τα αλλιεύματα. Εμείς λέμε ότι α, τα αλλιεύματα είναι, ανέρχονται σε τόσα, σε χ. Τι είδου συμφωνία είναι αυτή. Άρα τα νησιά του Σολομώντα δεν μπορούν να πιστοποιήσουν. Και ο μηχανισμός μπορεί να οδηγήσει και σε διαφθορά. Άρα κάποιος από τη δημόσια διοίκηση μπορεί να προωθήσει μια συμφωνία αλίας ...στη στιγμή που δεν υπάρχουν διαφανή στοιχεία για τα αλλιεύματα τα χρήματα ε, αποτελούν ψυχία χορηγήσεων, και, αλλά συμφώνησαν τα νησιά του Σολομόντα, άρα θα πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε πού έγινε η διαφάνεια. Η τοπική κυβέρνηση θα πρέπει να λογοδοτήσει για να βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης των ε, ντόπιων αλλιέων. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ε, αλλιεύματα σε τοπικό επίπεδο και εμείς ε, λαμβάνουμε όλο το κέρδος. θα πρέπει να ορίσουμε ελάχιστους όρους ε, που θα πρέπει να τηρηθούν σε περιφερειακό επίπεδο και επίσης να υπάρχει σε ταυτά χρονικά ε, διαστήματα μία εποπτεία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αρσένη με τις δύο τροπολογίες που υπέβαλε και τις οποίες υποστηρίζω. Υπάρχουν σχόλια συνάδελφοι. Ε, thank you very much. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ πολύ και για αυτή τη γνωμοδότηση για την αλληλευτική Συμφωνία. Επειδή συμμετέχω και στην Επιτροπή Αλίας, γνωρίζω πολύ καλά αυτές τις οικονομικές ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης και υποστηρίζω την ε, γνώμη σας. Επίσης διάβασα την αξιολόγηση της συμφωνίας ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και νήσων του Σολομόντα και το 35% των ποσών που καταβάλα του ποσού που καταβάλλονται προς τα νησιά του Σολομόντα η, μεταβαίνει προς υποστήριξη των ε, τοπικών πολιτικών. Αυτή, αυτό είναι το αναπτυξιακό σκέλος της αλλιευτικής συμφωνίας. Γι' αυτό μιλάμε και για αλλιευτικές εταιρικέ συμφωνίες. Και σύμφωνα με τη σύνοψη της αξιολόγησης, ως προς αυτό το σημείο, μάλλον η αξιολόγηση αναφέρει ρητά ότι το εταιρικό ε, σκέλος έχει αποτύχει. Και πέρα από τη συμφωνία, η Κοινή Επιτροπή ποτέ δεν μπόρεσε να συνέλθει από την απαρχή του πρωτοκόλου και δεν ορίστηκαν οι επιμέρους συνιστώσεις στα πλαίσια της εταιρικής συμφωνίας για τις αλλιευτικές ε, πρακτικές και τις ευρωπαϊκές επενδύσεις. Άρα αναφέρεται ρητά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε καν συναντήθηκε με εκπροσώπους των νήσων του Σολομόντα, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι το 35% προωθείται για τη βιώσιμη αλία στα νησιά του Σολομόντα και για να υποστηριχθεί ο εγχώριος τομέας αλίας. Υπάρχουν και πολλοί άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία σε αυτή την αποτίμηση για την οικονομία των νήσων. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα υποανάπτυκτη χώρα και ένα 14% ε, των πόρων προέρχονται από την Αλία. Άρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρίσκεται σε ένα πολύ πλούσιο τμήμα των ωκεανών. Άρα αυτή η χώρα θα πρέπει να διευρύνει την αλληλευτική της πολιτική. Όμως η αξιολόγηση λέει ότι δεν υπάρχει καν σχέδιο για το πώς θα πρέπει να εφαρμοστεί το εταιρικό σκέλος της συμφωνίας, αλλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε που άρχισε τη διαδικασία ούτε καν ε, συναντήθηκε με εκπροσώπους των νήσων. Αυτό είναι σκανδαλώδες. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μία διμερή συνάντηση καθώς και τεχνικές ομάδες που θα πρέπει να συνέλθουν, αλλά τα τέσσερα αυτά χρόνια είχαμε μόνο μία ε, τεχνική υφής ε, συνεδρίαση είναι σκανδαλώδες και αυτό είναι το ελάχιστο που μπορεί να υποθεί. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη σωστή πορεία με βάση τη διατύπωση. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει προσωπικό εκεί, γιατί έχουμε και το Κυριμπάτι και άλλες χώρες νήσους. Αν λοιπόν θέλουμε να προωθήσουμε αυτές τις εταιρικέ συμφωνίες θα πρέπει να είναι ουσιαστικές, να προωθήσουν την ανάπτυξη και τη βιώσιμη αλία σε αυτή την περιφέρεια του κόσμου και θα πρέπει να φροντίσουμε την εφαρμογή, δηλαδή ε, υποστηρίζω την αποτίμηση ότι θα πρέπει να υπάρχει προσωπικό από την Ευρώπη το οποίο να εγκατασταθεί εκεί. Επίσης, θα πρέπει να γίνει μια ενδελεχής αποτίμηση των πραγματικών αναγκών της χώρας. Δεν μπορούμε να χορηγούμε βοήθεια και μετά να ε, καταβάλουμε ένα αντίτιμο χωρίς να γίνει μια ενδελεχής ανάλυση της ουσίας, του περιεχομένου αυτής της οικονομικής εταιρικής σχέσης. Η αξιολόγηση αναφέρει ότι θα πρέπει να δοθεί συνέχεια από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί θα πρέπει να υπάρχει μία πλαισίωση για ένα πολιτικό διάλογο με τα νησιά του Σολομόντα. Εάν εφαρμόσουμε όλα αυτά που τόνισε ο εισηγητής Ντέβα, θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε μια ελευθερική συμφωνία αν είναι ε, πλήρως διαυγής και ε, αν αλλιεύουμε για το πλεόνασμα αλλιεύματος που δεν χρησιμοποιούν οι ντόπιοι. Αυτό αφορά και το δίκαιο της θαλάσσης των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχουν τέσσερα είδη σε αυτή την περιοχή. Το ένα είναι το skipjack και δεν έχουμε πρόβλημα με τα αποθέματα αλλά υπάρχει ο ερυθρός ο... που βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση διότι υπεραλλιεύεται και αυτό αφορά και το Big Eye Tuna, το μεγαλόφθαλμο τόνο που κινδυνεύει να υπεραλλιευθεί επίσης. Δεν υπάρχει ένα ανώτατο όριο αλλιευμάτων. Άρα δεν συμβαδίζουμε με τον νόμο που ορίζει για την αλίευση των πλεονασμάτων τόνου. Άρα καταρρεί το σύστημα σε σχέση με τον ερυθρό τόνο. Υπάρχουν ορισμένα αυστήρα κριτήρια που υποστηρίζουμε εμείς οι πράσινοι. Δεν είμαστε κατά των αλλιευτικών συμφωνιών εάν υπάρχουν ε, συμφωνίες οικονομικής εταιρικής ε, σχέσης και εάν αλλιεύουμε τα πλεονάσματα, τότε θα μπορούσαμε να χορηγήσουμε κονδύλια σε, αυτά τα, σε αυτές τις περιφέρειες του κόσμου. Και θα πρέπει να έχουμε μια περιφερειακή προσέγγιση, καθώς και την πολιτική πλαισίωση, τη σωστή πολιτική πλαισίωση. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι η παρούσα συμφωνία πλήρει αυτούς τους όρους. Καθόλου μάλιστα. Και αυτό είναι σκανδαλώδες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κυρία Λοβίν. Πολύ χρήσιμη αυτή η παρουσίαση που κάνατε και οι προτάσεις σας. Αν έλεγα ότι θέλω να αγοράσω αυτό για 65 ευρώ και το πουλάω 35.000 ευρώ μετά. Αυτό ισοδυναμεί με την τωρινή κατάσταση. Κάποιο πληρώνει 65 ευρώ για κάτι και το μεταπολεί ε, για 35.000 ευρώ. Ε, δηλαδή είναι κατάφορη ε, εκμετάλλευση αυτό που συμβαίνει. Όποιος δέχτηκε αυτό το πράγμα στα νησιά του Σολομωτά θα πρέπει να μπει φυλακή. Ε, ε, μας ζήτησε το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Αντρέας Φωτάνα πρώτος θα πάρει το λόγο. Κύριε Σιγητά, δεν είμαι ο Αντρέα Φοντά, ε, Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου λέγομαι. Εγώ είμαι τμήματάρχης και αποφάσισα να έρθω σήμερα ούτω ώστε να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας και με τους αξιότιμους βουλευτές τη Επιτροπή σας. Επιτρέψτε μου, αν έχουμε χρόνο, να σας κάνω μία σύντομη παρουσίαση για το νέο πρωτόκολλο και κατόπιν να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για ε, σχόλια που κάνατε εσείς και η κυρία Λεβίν. Ε, εξάλλου, η Ρίστα Εμπαρόδο ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα σχόλια της κυρίας Λεβίν. Λοιπόν, θα ήθελα να σκιαγραφίσω αδρά αυτό το νέο πρωτόκολλο, αρχίζοντας την παρέμβασή μου. Σε σχέση με το προηγούμενο πρωτόκολλο, κανονικά ε, ε, έχουμε κάνει ένα ποιοτικό άλμα στο νέο πρωτόκολλο. Ε, πάντως αναγνωρίζουμε δυστυχώς ότι δεν έχει λειτουργήσει σωστά ε, το πρωτόκολλο αυτό για διάφορους λόγους. Ε, αυτό το πρωτόκολλο ανήκει στο ευρύτερο πλαίσιο των συμφωνιών που έχει κλείσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με χώρες του Ειρηνικού Ωκεανού. Ε, με το Κυριμπάς έχουμε μια συμφωνία, με τη Μικρονησία άλλη μία ε, που ανανεώσαμε εσχάτως και Τέλος έχουμε αυτή τη συμφωνία με τα νησιά ε, solo model, δηλαδή έχουμε τρεις ε, συμφωνίες συνολικά, αλλά καθοριστική σημασία ε, για τον τόνο, διότι σε αυτή την περιοχή, στον Ειρηνικό ωκεανό, υπάρχει ένα πελώριο απόθεμα τόνου. Και άρα πρέπει να ε, είμαστε παρόντες στην περιοχή, όχι μόνο για να ε, ε, εκμεταλλευτούμε τα αποθέματα, αλλά και για να κατοχυρώσουμε μια αρμονική ανάπτυξη στον τομέα αυτά. Κατά τα λοιπά θα γνωρίζετε σίγουρα, κύριε Σιγήτα, ότι ο ευρωπαϊκός στόλος, ο αλλιευτικός στόλος δεν είναι ο μοναδικός που αλλιεύει σε αυτά τα νερά. Έχουμε ε, τέσσερις στράτες ε, εμείς ε, από ευρωπαϊκής πλευράς και άλλες χώρες αλληλείς μεγάλες έχουν ολόκληρες αρμάδες στο, στην περιοχή αυτή. Εμείς έχουμε μόνο τέσσερα τον αλλιευτικά. Αυτά για να γνωρίσετε τις διαστάσεις του προβλήματος. Βάσει του νέου πρωτοκόλλου προβλέπεται ε, το οικονομικό αντιστάθμισμα σε μεγάλο βαθμό να χορηγείται ε, στην ε, τομεακή αναπτυξιακή πολιτική. Και επανέρχομαι λοιπόν σε αυτά που ακούστηκαν για την εταιρική σχέση. Δεν περιορίζεται μια εταιρική σχέση στο να αλλιεύουμε κάπου και στη συνέχεια να αποχωρούμε. Η εταιρική σχέση έχει λόγο ύπαρξης μόνο Εάν με την συμφωνία χάρη στη συμφωνία αποδίδουμε μια δυναμική στον εγχώριο αλλιευτικό τομέα σε τρίτες χώρες, στη συγκεκριμένη περίπτωση στα νησιά του Σολομόντε, που για διάφορους λόγους ε, ιστορικούς, ε, κοινωνικούς, οικονομικούς δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί στο παρελθόν. Είναι ευκταίο λοιπόν να αναπτυχθεί ο τομέας και ο Επίτροπός μας αυτό επιθυμεί. Επιθυμεί να ακολουθήσουμε αυτή τη ρότα ώστε η συμφωνία να έχει θετικές επιπτώσεις ως προς την ανάπτυξη της τομεακής πολιτικής, της αλευτικής πολιτικής δηλαδή, σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή του κόσμου και πιο συγκεκριμένα στα νησιά ε, του Σολομόντα. Με την εταιρική σχέση λοιπόν έχουμε θετικά αποτελέσματα. Εσείς κάνετε μια απογραφή και εσείς και η κυρία Λοβίν. Ε, που ε, δεν είναι ε, ικανοποιητική. Πόρο απέχουμε από το να φτάσουμε σε ικανοποιητικό επίπεδο και δυστυχώς θα πρέπει να συμφωνήσουμε. Λοιπόν, αυτό το πρωτόκολλο καλύπτει μία τριετή περίοδο και προσφέρει αλλιευτικές ικανότητες που αποτιμώνται ως προς την πρόσβαση στα ύδατα. Πρόσβαση στην αποκλειστική οικονομική ζώνη των ίσων Σολομώντα λοιπόν για την αλλίευση του τόνου. Η πρόσβαση αυτή προσφέρεται σε τέσσερα τόνα αλλιευτικά που φέρουν ε, ε, σημαίνει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σύστημα των, ε, των αλλιευτικών συμφωνιών που ε, θα αναθεωρηθούν, έτσι, ρίστο εμπαρόδο, αυτό μας προβληματίζει στις υπηρεσίες μας, ε, αναρωτιόμαστε δηλαδή ποια πρέπει να είναι η βάση λειτουργία των, των αλλιευτικών συμφωνιών, αλλά πώ έχουν τώρα τα πράγματα σε κάθε περίπτωση, διότι ακόμη δεν έχει περατωθεί η μεταρρύθμιση, δεν έχει εγκριθεί. Το σύστημα λοιπόν είναι λίγαν απλό ο προϋπολογισμός της Ένωσης συμβάλλει σε ύψος 65% και πλειοκτείται πλειοκτήτες κατά 35% για το κόστος που πρέπει να καταβάλουμε για να κατοχυρώσουμε δικαιώματα πρόσβασης στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Για να υπολογίσουμε το, το, το, κόστος έχουμε και μια χωρητικότητα αναφοράς που προσδιορίζεται. Το τονάζ δηλαδή. Είπανε κάποιοι ότι αυτή η χωρητικότητα αναφοράς ε, δεν είναι ένα περιοριστικό ανώτατο όριο. Το δέχομαι αυτό. Ε, είναι γεγονός αυτό που αναφέρατε. Πλην όμω ε, θα διαπιστώσετε ότι από, από πρωτόκολλο σε πρωτόκολλο, από διαπραγματεύσει σε διαπραγματεύσει, επιχειρούμε να λαμβάνουμε υπόψη, όταν προσδιορίζουμε αυτό τη χωρητικότητα αναφορά, να λαμβάνουμε λοιπόν υπόψη το τωρινό επίπεδο αλλιευμάτων. Ε, και την κατάσταση του αποθέματος. Αν συγκρίνουμε λοιπόν το νέο πρωτόκολλο ε, που, διαπραγματεύτηκε τώρα, που διαπραγματευτήκαμε τώρα, αν το συγκρίνουμε με το παλιό πρωτόκολλο, θα διαπιστώσετε μείωση κατά ε, 6.000, από 6.000 μέχρι 4.000 τόνους σε σχέση με την χωρητικότητα αναφοράς. Για διάφορους λόγους κάναμε αυτή την αλλαγή και κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τις ε, επιστημονικές συστάσεις ε, του Περιφερειακού Αλλιευτικού Οργανισμού που καλύπτει την περιοχή του Ειρηνικού, δηλαδή το WCPFC που είναι ο, οργανισμ... ο περιφερειακός αρμόδιος οργανισμός που προφανώς είναι, όπου, συγγνώμη, είναι συμβαλόμενο μέρος ε, ε, τα νησιά του Σολομώντας. Τα πλαίσια αυτής της εταιρική συμφωνίας ε, πρώτη θέμεθα να συνεργαστούμε με τις τοπικές αρχές με στόχο να κάνουμε κοινέ πιλωτικέ εκστρατείε. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο που δεν υπήρχε στο προηγούμενο πρωτόκολλο και συμφωνώ απολύτως με τα σχόλιά σας ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις σχέσεις με αφενό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφετέρου τα νησιά του Σολομόντα. Ε, μιλήσατε για το σκάνδαλο, δηλαδή ότι η Μικτή Επιτροπή δυστυχώς δεν ε, μπόρεσε να συνεδριάσει τα τελευταία τρία χρόνια. Εγώ προσωπικά ε, θορυβήθηκα εξίσου ε, που το διαπίστωσα και σας διαβεβαιώ από τότε που επιτελώ αυτά τα καθήκοντά μου εδώ και έξι μήνες περίπου ε, προσπαθώ να ε, προωθήσω μια προσέγγιση που βασίζεται πολύ περισσότερο σε συνένεση ε, με τις χώρες με τις οποίες έχουμε συνάψει τέτοιες συμφωνίες, γιατί είναι θέμα αξιοπιστίας όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερο. Αυτές ε, οι συζητήσεις όπως η σημερινή, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να μας βοηθήσουν τόσο ώστε να το κάνουμε αυτό το ποιοτικό άλμα στο οποίο όλοι αποσκοπούμε, ε, το ποιοτικό άλμα στο οποίο αποσκοπεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διορθώσει τις ατέλειες του παρελθόντος. Ε, τώρα θα ήθελα να σας μιλήσω για κάποια βασικά στοιχεία, κάποια βασικά σημεία για να σας καταδείξω ότι παρά τις ατέλειες, παρά τα προβλήματα, ε, έχουν σημειωθεί κάποιες βελτιώσεις στο νέο πρωτόκολλο. Πιο συγκεκριμένα, ε, Κάποιοι μπορεί να κρίνουν βέβαια ότι είναι ανεπαρκές αυτό το στοιχείο, αλλά παρόλα αυτά, παρόλα αυτά ε, Έχουμε μία ρήτρα η οποία αξίζει μόνο και μόνο επειδή υπάρχει μία ρήτρα αναθεώρηση, ούτω ώστε η αδίποτε στιγμή αν διαπιστώσουμε παρατυπία να αναθεωρήσουμε το πρωτόκολλο ή αν εκτροχιαστούμε σχέση με τον αρχικό στόχο του πρωτοκόλλου. Δεν υπήρχε αυτό στην προηγούμενη συμφωνία. Εάν λοιπόν από οποιαδήποτε πλευρά ε, ελοχεύει κάποιο ε, κίνδυνο σε παρατυπία σε σχέση με τη συμφωνία υπάρχει η ρήτρα αναθεώρηση. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο διότι ε, ε, εδώ ε, χειριζόμαστε χρήματα φορολογουμένων εφόσον χρησιμοποιούμε τον κοινοτικό προϋπολογισμό και προφανώς τροφοδοτείται ο κοινοτικός προϋπολογισμός από τα χρήματα φορολογουμένων. Λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα αναστολής της εφαρμογής του, της συμφωνίας ή να θεωρήσουμε το κομμάτι σε σχέση με τη χρηματοοικονομική εισφορά, εάν ε, ε, ο στόχος της ε, τομεακής αναπτυξιακής πολιτικής δεν επιτευχθεί. Πρόκειται εδώ για βασική μεταρρύθμιση σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα. Η μεταρρύθμιση αυτή θα υλοποιηθεί και ανήκει στο οπλοστάσιο που ε, θέλουμε να συγκροτήσουμε με την επόμενη μεταρρύθμιση, ώστε να υπάρχει καλύτερη παρακολούθηση, συνενετική όμως παρακολούθηση, ε, ανάμεσα στα δύο συμβαλόμενα μέρη. Ε, λοιπόν, αισθητή είναι αυτή η βελτίωση που επιφέραμε στο πρωτόκολλο. Κατόπιν, θέλουμε να τονίσουμε την άμεση σχέση που πρέπει να υπάρχει με τις επιστημονικές γνώσεις, με τις επιστημονικές εγνωμοδοτήσεις και συστάσεις. Ε, θέλουμε να ενισχύσουμε έτσι περαιτέρω τη συνεργασία με τους επιστήμονες, ε, ακόμη και αν για τα μεταναστευτικά είδη η συνεργασία δεν είναι αποκλειστικά και μόνο συνάρτηση των επιστημονικών γνώσεων που έχουμε για τη συγκεκριμένη αποκλειστική οικονομική ζώνη, γιατί όπως, όπως λέει και το όνομά τους είναι μεταναστευτικά τα είδη και μετακινούνται από τη μία ζώνη στην άλλη και περνάνε από το ανοιχτό πέλαγος ε, για ε, ε, να φτάσουν στην επόμενη ζώνη. Οπότε πρέπει να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τις τεκμηριωμένες επιστημονικές συστάσεις που εκπονούν οι περιφερειακοί αλληλευτικοί οργανισμοί και συγκεκριμένα η WCPFC που είναι ένας περιφερειακός αλληλευτικός οργανισμός. Δεν θυμάμαι τώρα το, το, το, στα γαλλικά, δεν πειράζει, έχω κι εγώ ένα κενό μνήμης. Τελευταίο στοιχείο, κύριε Σίγητα. Έχουμε προβλέψει διατάξεις ως προς την κοινωνική ρήτρα για την επιβίβαση των ε, ναυτικών. Ε, κατελάχιστο όριο 25% ναυτικών που προέρχονται από χώρες και ε, αυτή είναι μια σημαντική περιφερειακή διάσταση και αποδίδουμε προτεραιότητα στους ε, αλληλείς που προέρχονται από τις νήσους Σολομόντα και προβλέπουμε την, ε, ε, μια συμβολή στο πρόγραμμα των παρατηρητών. Οι παρατηρητές είναι ένα ε, πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Πρόκειται για τους παρατηρητές που επιβιβάζονται στα αλλιευτικά κοινοτικά σκάφη. Θα υπάρχουν και παρατηρητές λοιπόν από, τους, από τα νησιά του Σολομόντα, πέρα από τους αλλιείς. Κάτι άλλο τώρα που δεν συνιστά νέο στοιχείο, αναφερόμαστε ε, στις ε, συμβάσεις ε, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για τους μισθούς, για τις συμβάσεις εργασίας και για την προστασία που πρέπει να κατοχυρώνεται. Ανοίγω και εδώ μια παρένθεση στο παρελθόν, πριν από μια εικοσαετία Φερρυπίν δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά και ε, συμφωνώ που χαρακτηρίσατε σκανδαλό την κατάσταση. Ε, ήταν σκανδαλώδη πριν από μία αιτία. Ήταν απαράδεκτη. Ε, τούτου λεξέντο και κλείνω την παρένθεση. Θα ήθελα να να σχολιάσω κάποιες παρατηρήσεις της κυρίας Λοβίν. Ε, με την οποία είχα την ευκαιρία να συναντηθώ πριν από δύο-τρεις μήνες σε ένα σεμινάριο που έγινε για το μέλλον της μεταρρύθμισης. Ήταν μια πρώτη ανταλλαγή που κάναμε, λίγα χρήσιμη και βλέπω ότι με πάθος ε, υπερασπίζεται ε, αρχές που με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο. Ε, πιστεύουμε πως εάν θέλουμε να αναπτύξουμε τις διμερείς σχέσεις μας με τις τρίτες χώρες ε, θα πρέπει να ε, κατοχυρώσουμε μόνιμη τακτική επαφή. Η κατάσταση στην οποία αναφερθήκατε κύριε Σιγητά και στην οποία αναφέρθηκε και η κυρία Λεβίν είναι απαράδεκτη. Δηλαδή το να μην συνεδριάζει η Μικτή Επιτροπή. βέβαια, ας μην υπερβάλλουμε γιατί η ε, για να συνεδριάσει η Μεικτή Επιτροπή πρέπει και τα δύο μέρη να ε, παρίστανται. Ε, για να γίνει αυτή η διμερή συνάντηση θα πρέπει ένα από τα δύο μέρη να το ζητήσει. Πλην όμως για διάφορα ζητήματα υπάρχουν κολλήματα, ίσως οικονομικής φύσης. Ε, δύσκολα λοιπόν μπορούμε να πείσουμε την τρίτη χώρα. Είναι άνθρωποι που έρχονται από την Ειρηνικό Είναι πάρα πολύ μακριά και κοστίζει πολύ ακριβά το ταξίδι. Δυσκολευόμαστε λοιπόν να τους πείσουμε να έρθουν να συζητήσουν μαζί μας ε, παρά τις ε, σχετικές διατάξεις της συμφωνίας. Εσχάτως όμως αναλάβαμε πρωτοβουλίες, δηλαδή ε, ε, συγκαλέσαμε μια συνεδρίαση στην αντιπροσωπεία που έχουμε στα νησιά Φίτζι, που είναι πολύ πιο κοντά στα νησιά του Σολομόντα παρά να έρθουν ε, μέχρι την Ευρώπη. Και επίση μια άλλη πρωτοβουλία που αναλάβαμε, τέλος πάντων είναι μια μικρή λεπτομέρεια, αποφασίσαμε να καλύψουμε τα οδηπορικά για κάποιου από αυτού του εμπειρογνώμονε για να μην υπάρχει αυτό το οικονομικό κόλλημα. Αποφασίσαμε να τους καλύψουμε τα οδηπορικά έξοδα. Ε, συμφωνώ πάντως ότι πρέπει να υπάρχει η τακτική επαφή και να τηρούμε τι διατάξει του πρωτοκόλου. Μία συνεδρίαση τη Μικτής επιτροπή. Ε, επιβάλλεται η συνεδρίαση τη Μικτής Επιτροπής, ε, διότι ε, θα πρέπει να από κοινού να γίνεται η αξιολόγηση της υλοποίηση ε, της ε, συμφωνίας ε, και συγκεκριμένα της διάστασης που άπτεται της τομεακής πολιτικής. Χωρίς συνεδρίαση, αν εφανταλλαγής απόψεων, δύσκολα μπορεί να λειτουργήσει το πρωτόκολλο. Λοιπόν, ναι, συμφωνώ για την συνεδρίαση, για αυτά που είπατε για τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Όπως είπε η κυρία Λοβίν, αυτή η συμφωνία παρά τις ατέλειες που ε, μπορούν να τις προσάψουν διάφοροι, επιτρέπει να ενισχυθεί ο πολιτικός διάλογος και επιτρέπει να δραστηριοποιηθούμε εντονότερα στην περιοχή. Λοιπόν, ξέρω ότι μακρηγόρησα, αλλά νομίζω ότι χρειαζόταν. Ναι, ζητώ συγγνώμη. Uh, Ευχαριστώ για, για αυτή την παρουσίαση, κύριε Αλεξάνδρου. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε μαζί μου σχετικώς με τη σκανδαλώδη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και χαιρετίζω την ιδέα ότι θα είσαστε η νέα σκούπα η οποία θα καθαρίσει το τοπίο και ελπίζω ότι στο μέλλον θα υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια. just, a uh, uh, Πολύ σύντομα. Κύριε Ντέβα, μιλάτε για 65 ε, ε, ευρώ τον τόνο για τον, ε, το ψάρι τόνο, αλλά ξέρετε ότι πληρώνουν ακόμη φθηνότερα εντό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δηλαδή 35 ευρώ τον τόνο, λοιπόν δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν πληρώνουμε το, για να πηγαίνουν στην άλλη άκρη του κόσμου να ψαρεύουν τόνο όταν δεν έχουμε χρήματα για να πληρώσουμε τα αεροπορικά τους εισιτήρια για, τις, ε, για τα νησιά του Σολομόντος. Ελπίζω ότι ο κύριος Αλεξάνδρου θα επανέλθει ή θα μου γράψει για να μου πει ποιος επωφελείται από αυτή την κατάσταση. Ποιος κερδοσκοπεί μάλλον. Διότι αν αγοράζετε ένα τόνο, τόνο 65 ευρώ και το πουλάτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 35.000 ευρώ θα πρέπει να ο καταναλωτής ε, ο οποίος έχει καταβάλει τη διαφορά να γνωρίζει ποιος ε, εποφελείται. Υπάρχει φορολογία, ε, τι, τι οφείλεται, διότι είναι ένα τεράστιο περιθώριο κέντρου στο οποίο είναι καθαρή εκμετάλλευση. Θα ήθελα λοιπόν είτε επισήμως είτε ατύπως γραπτός να μου πείτε ποιος ε, συγκεντρώνει αυτά τα χρήματα, αν τα κέρδη αυτά καταγράφονται και φορολογούνται εάν εξαφανίζονται στη φύση. Γενικώ θα ήθελα να ξέρω πώς αυξάνεται η αξία και ε, πού πηγαίνει. Ευχαριστώ. Ίσως στην επιστροφή αυτή, ε, με συγχωρείτε γιατί ήρθα τώρα, αλλά εφόσον θα συγγράψετε αυτή την ε, επιστολή, καλό θα ήταν να γνωρίζουμε, εφόσον το συζητήσαμε νωρίτερα, πόσο σημαντικό είναι να ενισχύσουμε τα κοινοβούλια στις ε, χώρες και να μας πείτε πώς θα περιλάβετε το κοινοβούλιο των νήσων του Σολομώντα και άλλες οργανώσεις ή της ε, τη συζήτηση για την κατάρτιση αυτής της ε, συμφωνίας αλληλείας και συνεργασίας και θα θέλαμε να καλέσουμε κάποιον από τις νήσους Σολομώντας σε αυτή την Επιτροπή για να δούμε όντως ποια είναι η επίπτωση εφόσον πρόκειται να υπάρξει μία αναθεώρηση και να πούμε αν συνενούμε ή όχι καλό θα ήταν ε, να έρθει κάποιος από την περιοχή εδώ Πολύ καλή ιδέα, περιμένουμε την επιστολή σας, διαφορετικά θα καθέσω το ερώτημα στο Στρασβούργο προς τον Επίτροπο. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει, ποια είναι η αλυσίδα, γιατί συμβαίνουν αυτά, ποιος επωφελείται, ποιος ε, εκμεταλλεύεται και γιατί είναι κατά διάκριση της ε, ε, τρίτης ε, χώρας η οποία εμπλέκεται σε ποια τράπεζα θα καταβληθούν τα χρήματα. Λοιπόν, τα χρήματα αυτά τα οποία θαυματουργά πολλαπλασιάζονται σε εκατομμύρια θα θέλαμε να γνωρίζουμε με διαφάνεια τι συμβαίνει, να το εξηγήσουμε στον Ευρωπαίο φορολογούμενο και νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση τώρα ή να έχω γραπτό τα σχόλιά σας και ε, με ένα ε, έγγραφο να γνωρίσω τι γίνεται. Τώρα φτάνουμε στη στιγμή της μπανάνας. Αύριο βέβαια θα είναι η ψηφοφορία επί του θέματος. Το επόμενο θέμα είναι η τροπολογία του κανονισμού ο, ε, για θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης ανεπτυξιακής συνεργασίας δηλαδή ε, θα μιλήσουμε για τις ε, χώρες οι οποίες παράγουν μπανάνες, ε, χώρες ΑΚΕ και που έχουν επηρεαστεί δυσμενώς από τις πρόσφατες εξελίξεις των διατάξεων εμπορίου σχετικά με αυτή την πρώτη ύλη και που έχουν επιρροή στην οικονομία τους. Η Επιτροπή Αναπτύξεως θα γνωμοδοτήσει και ο εισηγητής είναι ο κύριος Γκέρενς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις και καμιά δεκαριά προτάσεις σχετικά με την έκθεση για τα συνοδευτικά μέτρα σχετικά με τις μπανάδες. Πρώτη διαπίστωση. Πρόκειται για την απάντηση σε μία εμπορική συμφωνία η οποία είχε συναυθεί μεταξύ των χωρών ΑΚΕ που εξάγουν μπανάνες με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία συνεχίζει να εφαρμόζει μία προτιμησιακή συμφωνία με τις χώρες ΑΚΕ διότι κατόπιν ε, των ε, εκδηλώσεων διαφωνίας από τους άλλους εξαγωγείς μπανανών προς ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχτηκε να μειώσει τους εισαγωγικούς δασμούς της μπανάνας για όποιον δεν χαίρει των προτιμησιακών προτιμήσεων από 165 σε 140. Πρέπει να σας πω ότι η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Αναπτύξεως πρέπει να αναλύσει αυτή τη συμφωνία σχετικά με τα μέτρα ε, συνοδείας της μπανάνες ε, που αναφέρονται στην αναπτυξιακή βοήθεια και που πρέπει να ψηφιστούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής και εισαγωγός μπανάνας. Η μπανάνα είναι μία πλήρη στροφή, πολύ ε, τη στρώμε ε, ε, ιδίω όσοι σαν και εμένα θεωρούν ότι δεν ε, πρέπει να απέχουν από αυτή τη χρήση. Υπάρχει λοιπόν μία προτιμησιακή πρόσβαση της μπανάνας στην Ευρώπη από τις χώρες ΑΚΕ και επίπτωση στις χώρες που βρίσκονται ε, σε άλλες περιοχές από τις οποίες εισάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε αυτή την ε, ε, συμφωνία συνοδευτικών μέτρων για την μπανάνα διότι τότε το δικαστήριο στα πλαίσια του ΠΟΕ για την ρύθμιση των διαφορών θα μας κατεδίκαζε. Ε, είναι λοιπόν ε, μια ανησυχία που μας θίγει όλους. Όσον αφορά τα συνοδευτικά μέτρα για την μπανάνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαπραγματευτεί μία συμφωνία με τις χώρες ΑΚΕ και προτείνεται να ληφθεί υπόψη στις αποζημιώσεις που δεν ονομάζονται έτσι, ονομάζονται συνοδευτικά μέτρα, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι αποζημίωση δεν, ε, δεν μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει διαφορετικά για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, για να προωθηθεί η διαφοροποίηση των χωρών που πλήττονται από τα νέα μέτρα και να προωθήσουμε την μακροοικονομική σταθερότητα. Θα πρέπει, εφόσον πρόκειται για 10 χώρες οι οποίες ε, θα υποφεληθούν από αυτά τα συνοδευτικά μέτρα και για λόγους ε, οικονομίας χώρου θα τις ε, ονομάσω MRB και θα πρέπει να διαπραγματευτούμε συμφωνίες με κάθε μία χώρα χωριστά. Ε, κατά τρόπον ώστε να ε, προωθηθεί η δημοσιονομική βοήθεια στον τομέα αυτό ή στα πλαίσια συμφωνίας με τις χώρες όπου δεν ισχύουν αυτές οι δύο μέθοδοι ή δεν μπορούν να ισχύσουν για προφανείς λόγους θα πρέπει να ε, χρησιμοποιήσουμε διαφορετική προσέγγιση. Θα πρέπει όμως να προγραμματίσουμε αυτές τις δαπάνες για μία τριετία και μέτρα πρέπει να ληφθούν ήδη και μάλιστα πολύ γρήγορα για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν μέχρι το 2013 διότι δεν υπάρχει ρήτρα διαφυγής οπότε αν τίποτα δεν ε, αλλάξει νομοθετικά η συμφωνία αυτή θα πρέπει να τελειώσει το τέλος του 2013 και το λέω υποθετικά γιατί ελπίζω ότι θα υπάρξει μία ανανέωση της ε, συμφωνίας εκτός και αν επιμείνουμε σε αυτό το θέμα αποζημιώσεως σε μία νέα μορφή συνεργασίας. Όσον αφορά την ε, πολιετή στρατηγική, μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η κατανομή των ε, ενισχύσεων στις χώρες αυτές ε, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από τη σημασία εξαγωγών της ε, μπανάνας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την οικονομία της χώρας και το επίπεδο της οικονομίας η οποία θα ενισχυθεί. Έρχομαι τώρα στις προτάσεις που έχει διατυπώσει η δικιά σας Επιτροπή και τις υποβάλλω προς ε, ε, ενημέρωση διότι έχω ζητήσει από την Επιτροπή να υιοθετήσει αυτές τις προτάσεις. Καταρχήν ε, τα μέτρα αυτά για την μπανάνα θα πρέπει να επηρεάσουν την συμφωνία ε, και τώρα αναφέρονται μόνο σε 1,5% της τελικής τιμής του προϊόντος πράγμα το οποίο ε, θυμίζει αυτά που είπαμε για την προηγούμενη έκθεση για τη σχέση της τιμής που πληρώνεται στην εξαγωγική χώρα σε σχέση με αυτήν η οποία πληρώνεται από τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Εδώ ε, πληρώνεται εις τον παραγωγό ΑΚΕ 1,5% της τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής στην Ευρώπη. Γι' αυτό και είχαμε ζητήσει μία μελέτη σχετικά με το δρομολόγιο της μπανάνας για να δούμε ποιος ε, ε, παίρνει τι κάθε φορά που αλλάζει η διοκτήτη μπανάνα αυτή. Είναι πολύ κακό το αποτέλεσμα. Ε, ε, μάλιστα αν μιλήσουμε απλώς ε, για κακό είμαστε πολύ μετριόφρονες και πρέπει να κοιτάξουμε πολύ κριτικά τις αδυναμίες της ανταμοιβή των παραγωγών στις χώρες παραγωγής μπανάνας. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη τα μέτρα της καταπολέμησης της στόχιας για να μπορέσει ε, όλη η σειρά που εμπλέκεται να ε, ικανοποιείται ε, επαρκώς θα πρέπει η εργασία να συνάδει με τις, εργασίες, με ε, διατάξεις του ΠΟΕ ε, και θα πρέπει και ο παραγωγός να ανταμείβεται διαφορετικά δεν αξίζουμε τίποτα σαν πολιτική θα πρέπει να υπάρχει και μια δίκαια καταμονομή των εισοδημάτων που προέρχονται από τις μπανάνες και το λέγω αυτό διότι μπορεί κανείς να εξασκεί πολιτική εις βάρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και όποτε χρειάζεται γίνεται στα πλαίσια της αναπτυξιακής βοήθειας η οποία καταναλύσχεται σε σχέση με το εσωτερικό ε, ΑΕΠ. Ε, υπάρχουν όμως και μέτρα που δεν μας κοστίζουν τίποτα και γι' αυτό έχω προτείνει και το τρίτο μέτρο που καλεί όλη την ε, αλυσίδα που εμπλέκεται στο εμπόριο των μπανανών να συμφωνήσει ως, το, ως προς το κοινό αποτέλεσμα και ε, να υπάρξει μία ενιαία πειθαρχία και αντιμετώπιση των παραγωγών μπανάνας. Είναι κάτι νέο το έχουμε κάνει όμως και σχετικά με την κρίση του γάλατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η παραγωγή γάλατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ικανοποιήθηκαν για τη τιμή την οποία ελάμβαναν και πέτυχαν να συζητήσουν με όλους αυτούς οι οποίοι, είναι, οι οποίοι εμπνέκονται στην διαδικασία από τον παραγωγό μέχρι τον τελικό καταναλωτή ε, και αυτό είχε μεγάλη απήχηση στην Ευρώπη γιατί λοιπόν να μην ε, εμπνευστούμε για να αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο την ανταμοιβή των παραγωγών μπανάνες. Μετά, όσον αφορά τις ε, συνδρομές και εδώ θα μπορούσαμε να αναφέρουμε διάφορα κριτήρια πάντοτε μιλάμε για ιστορικά κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη ε, όσον αφορά την δικλίδα κατανομής και ε, θα ήθελα να υποβάλω την ιδέα προσκέψη, δηλαδή εάν ερευνούμε υπερβολικά το παρελθόν, δεν ε, αξιολογούμε πλήρως ε, το πρόσφατο παρελθόν, τα τρία τελευταία χρόνια παραδείγματο χάρη. Τρίτον, ε, μηχανισμοί συντονισμού με άλλα ταμεία θα πρέπει να καταρτιστούν σχετικά με τις, τα συμπληρωματικά μέτρα διότι επιμένουμε εις ε, την ε, συνεκτικότητα της πολιτικής σε όλους τους τομείς, αλλά θα πρέπει ο ένας να ξέρει τι κάνει ο άλλος. Δηλαδή, αν τα κράτη-μέλη εμπλέκονται σε προγράμματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με ε, τα συνοδευτικά μέτρα δεν θα πρέπει να υπάρχουν επικαλύψεις ε, και οι επιπρόσθετες ε, σύνδρομες των κρατών μελών θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Κάθε δέσατη της χώρας μπορεί να ε, λάβουν υπόψη την αξιολόγηση που θα πρέπει ε, να λάβει υπόψη όλες τις συμφωνίες. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν δίκτες για στήριξη δημοσιονομική και νομίζω ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στο θέμα αυτό τα δε αποτελέσματα σχετικά με τη συγκεκριμένη αναθεώρηση στον τομέα των μπανανών θα πρέπει να γνωρίζουμε τι επιζητούμε και να αντικατοπτιστεί αυτό στο έγγραφο σε σχέση με, την α, κίνηση του προγράμματος ΕΡΑΜΠΕ και θα πρέπει να υπάρξει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και για τις χώρες που θα υποφεληθούν και ε, για τα θέματα που έχουν σχέση με τα φυτοφάρμακα, ε, τα ζυζανιοκτώνα. Σε αυτό θα ήθελα να απαντήσω στο σχόλιο των Πρασίνων στα πλαίσια αυτής της συζητήσεως ε, στην Επιτροπή μας. Αναφέρομαι στην αξιολόγηση και επιμένω, διότι Ακόμη και αν δεν επιτύχουμε να αξιολογήσουμε συστηματικά όλες τις συμφωνίες με τις 10 χώρες, με το φόβο του αστιφύλακα θα μπορέσουμε να επιτύχουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι να γνωρίζουν ότι ενδέχεται να υπάρξει έλεγχος και ε, ε, δεν θα πρέπει θα πρέπει να ε, φροντίσουμε να καλυφθεί η ψαλίδα αυτή των 190 μέχρι 210 ευρώ. Επίσης ε, θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση των εργαζομένων ε, επιτόπου γιατί πιστεύω ότι ο τομέας αυτός που είναι το αντικείμενο αυτής της εκθέσεως αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα διότι η Αφρική γενικώ και οι χώρες ΑΚΕ ε, ειδικότερα εξάγουν ένα προϊόν μια πρώτη ύλη με χαμηλή ε, αξία όπως ε, έχω επαναλάβει και θα πρέπει να διερευνήσουμε τις πίστες για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ε, αξιοποιήσουμε την τροποποίηση της μπανάνας απαρχής και να υπάρχει η δυνατότητα αναδιατάξεως των χώρων καλλιεργίας της μπανάνας, της μπανοφυτίας ε, είναι κάτι που πρέπει να το να ελέγξουμε και να μελετήσουμε ε, γιατί είναι κάτι που έχει σχέση με την αηφόρα ε, ανάπτυξη και εδώ έχουμε μία αρχή ε, την οποία έχει οθετήσει η Επιτροπή μας επί του θέματος, δηλαδή ότι τα μέτρα θα πρέπει να συνάδουν με τις δυνατότητες αφομοιώσεως των ε, χωρών, διότι όταν μιλάμε ε, για 190 εκατομμύρια ως δεσμεύσεις δεν πρόκειται για ουσιαστικές πληρωμές εάν στο τέλος δεν έχουν καταβληθεί τα 190 εκατομμύρια ή δεν μπόρεσαν να ε, δαπανηθούν ε, αυτό μπορεί να εξαρτάται και από τη δυνατότητα αφομοιώσεως ε, της εν λόγω χώρας και δεν θα πρέπει να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό εις βάρον των εργαζομένων μέσω εκτενούς χρήσεως ζυζανιοκτώνων και αυτό ίσως ε, σας φαίνεται ίσως ε, σαν ανεδαφικό, αλλά στις ε, εμπορικές συμφωνίες είμαστε η πρώτη επιτροπή που δεν μπορεί να αναφερθεί στην κατάσταση των τον, η οποία ισχύει στην πραγματικότητα διότι ε, ε, ένας συνδικαλιστής μου είπε ότι στο Μπαγκλαντές συγκεκριμένα κατόπιν ε, της απελευθερώσεως της αγοράς κλωστοϊφαντουργικών η εβδομαδιαία ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας έφτασε σε 72 ώρες. Οπότε, ποιος, ποιος αντιμετωπίζει αυτά τα απαράδεκτα θέματα και πώς θα λύνει. Το ίδιο νομίζω συμβαίνει και για τις βανάνες όπως και για τα κλωστοϊφαντουργικά και οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες στις χώρες μας είναι νομότυπες και καλούνται να προστατεύσουν τον καταναλωτή αλλά αν ε, και άρα δεν πρέπει να εκτίθενται ε, στα ζυζανιοκτώνα άνθρωποι, αλλά όταν δεν υπάρχει νομοθεσία στις χώρες επιτόπου κάνουν ό,τι τους ό,τι θέλουν. Οπότε γι' αυτό το λόγο αναφέρομαι, αλλά αυτό είναι το θέμα της μπανάνας, δηλαδή δεν είναι ένα περίπλοκο φρούτο, αλλά ό,τι έχει σχέση με αυτά τα φρούτα είναι πολύ περίπλοκα. Και η μελέτη την οποία ζητήσουμε τονίζει αυτό τον περίπλοκο χαρακτήρα γιατί αναφέρεστε σε όλα τα συστατικά στοιχεία αναπτύξεως όταν φύγετε αυτό το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και περιμένω τις πολυάριθμες ερωτήσεις άπαξ και η παρουσία έχει αυξηθεί από την αρχή της συνεδριάσεως βέβαια όχι τόση όσο εχθές το βράδυ μπροστά στις οθόνες του public viewing, αλλά τουλάχιστον σε σχέση με όσους παριστάντου στην αρχή της συνεδρίασης. Και θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να σας πω ότι είμαι ένας καλός σας φίλος. Ευχαριστούμε κύριε Γκέρενς. Πολύ χρήσιμη αυτή η παρουσίαση. Αναφερθήκατε στη μελέτη σας και είπατε ότι κάνατε και μία επιπρόσθετη μελέτη. Και αν κρίνουμε από τη τιμή που καταβάλει ο Ευρωπαίος πολίτης, ο παραγωγός κερδίζει ένα, ένα 0,51%. Θα ήθελα να ξέρουμε ποιοι είναι οι μεσάζοντες, τι κέρδη έχουν, ποιοι είναι αυτοί οι μεσάζοντες, πώς το καταφέρνουν. Γιατί εάν συνεχίσουμε το θέμα, ίσως να είμαστε σε ε, θέση να βγάλουμε αυτά τα χρήματα, να τα αφαιρέσουμε από τους μεσάζοντες μάλλον και να πάνε στους παραγωγούς. Για την αλία. Είπαμε ότι ο παραγωγός μπανάνας παίρνει 1,51% και τα νησιά του Σολομόντα παίρνουν το 0,19% της τελικής τιμής του τόνου. Δηλαδή μιλάμε για ακραία εκμετάλλευση και σε ευρεία κλίμακα. Ο κύριος Τυρολίων. Τυρολιά. Η πρόταση κανονισμού των υπηρεσιών της ε, Κομισιόν δεν είναι ικανοποιητική ούτε ως προς τον τύπο ούτε ως προς την ουσία. Όπως είπα στις προγενέστερες συζητήσεις μας, στον προϋπολογισμό του 2011, είναι δύσκολο για την Επιτροπή μας να δεχτεί την Επιτροπή Χρηματοδότησης, διότι πρόκειται για ένα νέο μέσο συνεργασίας. Επειδή ε, προέρχομαι από μία περιοχή του κόσμου που παράγει, που καλλιεργεί ε, μπανάνα και επειδή έχει πληγή θεωρώ ότι μπορώ να δεχτώ την αρχή πρόταση, αλλά δέχομαι την πρόταση Επιτροπής να ξαναχρησιμοποιήσει τα 57 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπονται για χρηματοδότηση δράσεων για την υγεία κατά πολέμηση της ε, λιτότητας, της πείνας μάλλον, και αυτές είναι προτεραιότητες για την Επιτροπή μας. Επί της ουσίας, ως προς τον τρόπο χρηματοδότησης, δηλαδή με βάση τους προγενέστερους κανονισμούς του 94 και 99 είδαμε ότι ένα μέρος των κονδυλίων όπως είχαν κατανεμηθεί χρησιμοποιήθηκαν πολύ καλά ιδιαίτερα με βάση τον κανονισμό του 99 τα προϊόντα, μάλλον τα επενδυτικά σχέδια που ήταν ολέθρια. Επειδή ήταν λιγότερο ανταγωνιστικές οι μπανάνες από τις χώρες και δυνάμει των αποφάσεων του ΠΟΕ, θα έπρεπε να δοθεί μία βοήθεια στους παραγωγούς ανάλογα με την ε, κατάσταση της αγοράς. Αλλά φαίνεται ότι αυτή δεν είναι η πρόταση που δέχεται η Κομισιόν. Ως προς τους ε, ε, τρόπους κατανομής για τις δέκα αυτές χώρες δεν είναι ο πιο διαφανής τρόπος. Εάν η Κομισιόν έλαβε υπόψη τρία κριτήρια, δεν φτάνουμε σε ένα συντελεστή στάθμισης έτσι ώστε οι χώρες να γνωρίζουν πόσα χρήματα διαθέτουν. Ενώ οι χώρες, οι αφρικανικές χώρες που λαμβάνουν αυτό το BAM έχουν μία δεκαετή περίοδο και με βάση την πρόταση της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν τους βοηθάει να φτάσουν σε μία ε, σωστή στρατηγική. Αναμένοντας ε, τις περαιτέρω εξελίξεις, αυτά είναι ορισμένα από τα σχόλια που θα ήθελα να προωθήσω. Είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε την άποψη της Γουαδελούπης σε σχέση με τους μπανανοπαραγωγούς. Ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ. Δέχομαι τις, ε, τα σχόλια του Πατρίς Τυρολιάν γιατί βλέπουμε ότι με βάση τα στοιχεία που μας έδωσε ο κύριος Γκέρενς φαίνεται ότι μας κατακλέβουν, γιατί θα πρέπει να βασιστούμε σε στοιχεία. Χαίρομαι με την προσέγγιση του κυρίου Γκέρενς σε σχέση με την ενδυνάμωση, την ενίσχυση των παραγωγών μπανάνας. Θα ήθελα να πω για τους παριστάμενους ότι υπόθηκε ότι αυτό το απλό φρούτο δεν είναι απλό φρούτο. Γιατί όταν μιλάμε για ορισμένα είδη σαλάτας, εξωτικές σαλάτες, ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι για ένα συστατικό που δεν είναι απλό φρούτο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλαπλώς. Δηλαδή, θα πρέπει να απαντήσει και η Κομισιόν και το Συμβούλιο για την κατάσταση όπως επικράτησε. Um, anybody else? Κάποιος άλλος. Η Κομισιόν. Ο κύριος Merci, Monsieur le Président, et merci au rapporteur, Monsieur Goerens, et aux autres intervenants. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες γιατί όπως είπε και ο κύριος Γκέρενς μιλάμε για πολλές αναπτυξιακές πτυχές έχει μεγάλη σημασία ο τομέας της μπανάνας για τις ε, άμεσα ενδιαφέρομενες χώρες. Καθίσταται σαφές ότι με βάση το μέσο συνεργασίας υπάρχουν όλα αυτά τα ε, στοιχεία τα οποία σχετίζονται και με αυτές τις αποστολές συνοριακής συνδρομής. Και υπάρχει και το περιβαλλοντικό προφίλ αυτό των 10 χωρών. Ο κανονισμός BAM προβλέπει ότι οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και να εντάσσονται στην στρατηγική στην αναπτυξιακή στρατηγική. Για να απαντήσω, θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για συνοδευτικά μέτρα. γιατί δεν πρόκειται για αντιστάθμιση, αλλά για συνοδευτικά μέτρα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της συμφωνίας. Όσον αφορά τα στοιχεία, το δίκτυο φτώχεια και το επίπεδο του 1,51% θα ήθελα να σας τονίσω ότι στα πλαίσια του αναπτυξιακού μέσου θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στη φτώχεια. Και αυτό το στοιχείο εδώ θα πρέπει να εγγραφεί. Θα ήθελα να πω ότι 1,5% της τιμής που καταβάλλεται από τον ε, Ευρωπαίο πολίτη ε, αποτελεί ένα εισόδημα που δεν είναι καθόλου αμεληταίο για τον εργαζόμενο. Βεβαίως αυτές οι καταστάσεις βρίσκονται σε ε, αυτές οι χώρες βρίσκονται σε μια κατάσταση ένδυας γενικότερα. Γι' αυτό θα πρέπει να στηρίξουμε το εισόδημά τους σε σχέση με τα θέματα που εφήγησαν για τις θετικές επιπτώσεις ως προς την αλυσίδα παραγωγής το 1,51% όπως μας είπε ο κύριος Γκέρενς και μιλάμε για μία δίκαιη κατανομή των εισοδημάτων που προέρχονται από την μπανάνα. Πιστεύω ότι το, ο μηχανισμός BAM είναι καταλήτης σε αυτή την ε, διεργασία. Με βάση, τον, ε, με βάση τις πολιετής ε, στρατηγικές υποστήριξης και όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στα πλαίσια ενός πολιτικού διαλόγου, έτσι ώστε αυτή η ε, συνοριακή συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το BAM, να ενταχθεί πλήρως σε αυτά τα πλαίσια. Ως προς την εφαρμογή του BAM υπάρχει μία αλληλεπίδραση όπως προβλέπεται με τους άμεσα εμπλεκόμενους και όταν γίνει μία συζήτηση για τις στρατηγικές υποστήριξης σε πολιετές πλαίσιο θα πρέπει όλα αυτά να ενταχθούν σε μία ευρύτερη στρατηγική. Άρα το BAM, το BAM είναι καταλήτη σε αυτά τα πλαίσια. Ως προς την κλίδα κατανομής, πιστεύουμε ότι τα τρία κριτήρια που υποβλήθηκαν είναι εξισορροπημένα και αποτελούν μια καλή εκτίμηση των αναγκών προσαρμογής κάθε χώρας. Τα δύο πρώτα κριτήρια σχετίζονται με την σημασία του εμπορίου μπανάνας ως μια κατόγκον παραγωγή στα πλαίσια του GNI και το τρίτο κριτήριο συγγνώμη, είναι το κριτήριο φτώχειας για να δούμε ποιος είναι ο αναπτυξιακός δείκτης. Και έχει μεγάλη σημασία στα πλαίσια της ε, φτώχειας ε, να δούμε ότι ε, πώς ακριβώς προσμετράται η φτώχεια, ποιος είναι ο δείκτης ένδυας, ο οποίος θα πρέπει να ενταχθεί εδώ, μέσα στα πλαίσια των ε, τριών κριτηρίων που αποτελούν μια καλή εξισορρόπηση μεταξύ των αναγκών προσαρμογής και της ε, αύξησης του αναπτυξιακού ρυθμού. Ως προς τα στοιχεία μπορώ να σας πω ότι θα πάμε πέντε χρόνια πίσω για τα στοιχεία που σχετίζονται με την κατανομή των ε, κριτηρίων αυτών. Ε, γίνονται ασκήσεις προσωμείωσης, αλλά είναι δύσκολο να δώσουμε οριστική μορφή σε αυτήν την εργασία τη στιγμή που η νομική βάση δεν έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Αυτή η ανάγκη σχετίζεται με το γεγονός ότι το ΜΠΑΜ είναι αναπόσπαστο τμήμα μίας σειράς μέτρων και υπάρχουν προβλήματα χρονισμού και για την ε, εφαρμογή αυτού του πλαισίου. ως προς τα κριτήρια. Στο σημείο 6 του κ. Γκέρνς μπορούμε να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα σχόλια και θα ληφθούν υπόψη στον αναπτυξιακό διάλογο με τις χώρες του τρίτου κόσμου. Όσον αφορά το θέμα των εργαζομένων και τα περιβαλλοντικά, ήδη απάντησα. Έχουμε πρόθεση να προωθήσουμε μια περιβαλλοντική αποτίμηση στα πλαίσια της κατάρτισης στρατηγικών υποστήριξης και οι 10 εμπλεκόμενες χώρες έχουν ένα περιβαλλοντικό προφίλ, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα θετικό. Οι περισσότερες ε, ενδιαφέρομενες χώρες έχουν ε, κυρώσει τη συνθήκη του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για την προστασία των εργαζομένων. Ε, ορισμένες χώρες έχουν κυρώσει μόνο ένα τμήμα αυτής της σύμβασης και ίσως το BAM, αυτή η αποστολή, η αποστολή συνοριακής συνδρομής, μπορεί να είναι καταλήτης και για τις ε, περαιτέρω κυρώσεις διότι οι χώρες θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή αυτές τις συμβάσεις αλλά το BAM, η αποστολή συνεργικής συνδρομής, μπορεί να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Ως προς τη μεταποίηση της μπανάνας, από όσο γνωρίζω, πρόκειται για μια δραστηριότητα που είναι αρκετά περιθωριακή στις ενδιαφερόμενες χώρες και στις χώρες παραγωγούς και είναι πολύ πιο ενδιαφέρον να προβάλλουμε τη μεταποίηση σε άλλα φρούτα που παράγονται πιο μαζικά και πιστεύουμε ότι στον τομέα της ε, μπανάνας δεν υπάρχουν μεγάλες διέξοδοι ε, στον τομέα της μεταποίησης διότι αυτό που μπορεί να προωθήσει κανείς κυρίως είναι το προϊόν όσο έχει στις αγορές. Σε σχέση με τις αξιολογήσεις και το monitoring, Γενικότερα θα ήθελα να πω σε σχέση ε, με τα σχόλια, με τα αρχικά σχόλια, τη στιγμή που δεν υπάρχει μελέτη αντικτύπου, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αποτιμήθηκε το προγενέστερο πρόγραμμα. Η έκθεση είναι διαθέσιμη με την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου Και Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να ενσωματώσουμε και το BAM. Ως προς τα αναπτυξιακά προγράμματα της Κομισιόν θα υπάρχει ένα πλαίσιο εποπτείας και μία μελέτη αντικτύπου που μπορεί να διενεργηθεί στο τέλος του προγράμματος. Αυτή η μελέτη αντικτύπου δεν μπορεί να γίνει το 2012-2013, διότι τότε θα τεθούν σε εφαρμογή αυτά τα προγράμματα. Πιο ρεαλιστικό θα ήταν να μιλάμε για 2015-2016. Ε, Ως προς την ε, δυνατότητα απορρόφησης των δικαιούχων, αυτό δεν μας απασχολεί είναι θέμα καλής ε, διαχείρισης και θα τελειώσω εδώ κύριε Πρόεδρε νομίζω. Σε σχέση λοιπόν με τα δύο ζητήματα, σε σχέση με το θέμα του προϋπολογισμού, η πρόταση της Κομισιόν βρίσκεται επί Βεβαίως υπάρχουν ορισμένα χρήματα που αφορούν την επαναχρηματοδότηση και αρχικά η Κομισιόν ήθελε να χρησιμοποιήσει τα δημοσιονομικά ε, περιθώρια που υπήρχαν. Υπάρχει και μία πρόταση ε, τροποποίησης του προϋπολογισμού. Μιλούσαμε για 25 εκατομμύρια τα οποία ήταν αναγκαία κατά την Κομισιόν να χρησιμοποιηθούν για την επαναχρησιμοποίηση τώρα πόρων για το 2010 ένα ε, μέρος αφορά έναν ευέλικτο μηχανισμό και ένα άλλο τμήμα αφορά την επαναχρησιμοποίηση του food facility. Σε ευχαριστώ και με συγχωρείτε που μακρηγόρησα. Σας ευχαριστούμε κύριε Ντύμπουα. Πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Δεν ε, μακρηγορήσατε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων για τον εισηγητή μας. Είναι πολύ ανοιχτός ο διάλογος που έχουμε και έτσι μπορούμε να συνδράμουμε στην ε, πόνηση της τελικής συμφωνίας με ουσιαστικό τρόπο. Κύριε Γκέρενς, ε, θα θέλατε να κάνετε κάποια καταληκτικά σχόλια, μήπως. Μα ήταν ε, εξαιρετικά εύστοχα τα σχόλια που κάνατε μετά την παρουσίασή μου. Στυλιτεύσατε το ποσοστό, το 1,5% που παίρνουν οι παραγωγοί και δικαίως. Θα ήθελα να ξέρω αν στον τομέα της μπανάνας μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Δεν κατηγορώ κανέναν, θέλω να ξέρω απλώς αν είναι δυνατόν. Λένε οι Αφρικάνοι, περίμενα να περάσεις ε, το ποτάμι για να πεις ότι είναι κακομούτσινοι οι κροκόδιλοι. Οπότε ας περιμένουμε να περάσουμε το ποτάμι, να δούμε ποιες είναι οι ανομαλίες ε, του συστήματος. Σας πειράζω λίγο, αλλά έτσι ήθελα να απαντήσω στα σχόλιά σας. Κύριε Τιεγολιά, η δημοσιονομική πλευρά που ε, έθιξε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, είναι σημαντική και χαρακτηρίζεται από αυτό που είπατε, από την χρήση 57 εκατομμυρίων ευρώ στα πλαίσια του DCI, του Οργάνου Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Ε, συγγνώμη, αλλά όλοι θα πρέπει να ε, μεριμνούμε ώστε να είναι συνεκτική η δράση μας, όχι μόνο εμείς. Ε, θα εξακριβώσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά δεν μπορείτε να μας κατηγορήσετε για έλλειψη συνοχής. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που επιδιώκουμε να είναι συνεκτικές οι δράσεις μας. Για τα κριτήρια ε, ομολογώ ότι δύσκολα, είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε ένα ορθό σετ κριτηρίων. Ε, κυρίως ε, για τη μορφή από ταμείευσης. Δεν ε, ισχύουν τα ίδια για όλους. Αυτές οι χώρες έχουν μικρότερες δυσκολίες ως προς την απορρόφηση των κονδυλίων, αλλά δυστυχώς όλοι όσοι λαμβάνουν τι επιδοτήσει μόνο μέσα από τα προγράμματα αντιμετωπίζουν σημαντικότατε δυσκολίε. Αυτό είναι θέμα διακυβέρνηση. και φυσικά πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση ώστε να υπάρχει σωστή χρήση των κονδυλίων. Κύριε Κάσμαν, ο σοσιαλιστής καλά κάνει και ακολουθεί τους φιλελευθέρους και ασχολείται με τα κοινωνικά πρότυπα και κυρίως με τα θεσμικά όργανα που εμπλέκονται. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας προφανώς έχει ρόλο να διαδραματίσει στον τομέα αυτό. Ε, στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες ε, προφανώς είναι ένας θεσμικός εταίρος και έχει πολύ χρήσιμη εμπειρία στον τομέα αυτό και πρέπει να συμβάλλει. Τώρα για το χαρακτήρα της μπανάνας. Εγώ είπα ότι φαίνεται απλό το φρούτο, αλλά είναι ε, περίπλοκο. Και εκείνο μου λέει ότι είναι εξωτικό το φρούτο, και, ε, το φρούτο και μετά μου λέει ότι είναι ερωτικό. Ε, δεν κατάλαβα το λογοπαίγνιο του κ. Κάσμαν. Αν μπορεί και έχει την καλοσύνη, μου το εξηγήσει. Ε, ως προς τις ε, παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, νομίζω ότι συμφωνούμε για τα σημαντικότατα στοιχεία. Αλλά υπάρχει μια παρανόηση, μια μικρή παρανόηση για την αξιολόγηση. Εγώ θέλω να γίνεται συστηματική αξιολόγηση των συμφωνιών με αυτές τις χώρες. Ή τουλάχιστον να προβλεφθεί η υποχρέωση και δυνατότητα να γίνεται η αξιολόγηση. Αυτό προϋποθέτει ότι η αξιολόγηση θα αποτελεί μέρος αναπόσπαστο κάθε προγράμματος που διαπραγματευόμαστε με κάθε μία από αυτές τις δέκα χώρες. Η όρια η αναφοράς θα πρέπει να είναι γνωστή από την έναρξη του προγράμματος. Γιατί πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς θα αξιολογήσουμε. Και αν η πολιτική μας προσανατολίζεται προς τα αποτελέσματά της, και ποια είναι τα αποτελέσματα, προφανώς η καταπολέμηση της ένδυας. Άρα η διαδικασία θα πρέπει να ε, λαμβάνει υπόψη αυτή την υποχρέωση παραγωγής αποτελεσμάτων. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να προσδιορίσουμε τους όρους διεξαγωγής της αξιολόγησης. Πώς να διαπιστώσετε πώς έχει η κατάσταση, πώς να αξιολογήσετε το, τον αντίκτυπο μετά το πέρας της διαδικασίας, αν δεν γνωρίζετε εξ αρχής ε, τους όρους αναφοράς, γιατί αλλιώς δεν θα είμαστε ουδέτεροι σε σχέση με την ακολουθητέα πολιτική. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ χρηστή αρχή για όλα, όλες τις δράσεις που προσανατολίζονται προς τα αποτελέσματα και κρίνονται βάσει των αποτελεσμάτων τους. Ε, έτσι νομίζω θα διαλύσουμε αυτή την παρανόηση που υπάρχει και θα, δεν θα ε, είμαστε ε, όμοιροι αυτού του διαλόγου κοφών. Πέραν αυτού δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Ο κύριος Κάσμαν μόνο να μας εξηγήσει το λογοπαίγνιό του. Θέλω, ζητώ διευκρινιστή τι ακριβώς εννοούσε ο κύριος Κάσμαν. Σας ε, ευχαριστώ και ελπίζω, δεν ξέρω, απάντησα σε όλους. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Γκέρενς, ε, δεν ξέρω αν μπορεί να εξηγήσει ο κύριος Κάσμαν ή αν πρέπει στις 30 ε, Αυγούστου θα γίνει η συζήτηση και στις 15 Σεπτεμβρίου η ημερομηνία, η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Σας ευχαριστώ όλους όσους ε, συμμετείχατε στη συζήτηση και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρενέβη. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Προστασία της βιοπικιλότητας ε, για και ε, ανάπτυξη συστημάτων για την εκπλήρωση των στόχων της χιλιετίας. Το 2010 είναι η χρονιά της βιοπικιλότητας, στην ανακήρυξη ΟΗΕ, Στη χρονιά βιοπικιλότητας. Το 2002 έγινε Παγκόσμια Σύνοδος στο Ιωάννησμπουργκ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατέληξαν ε, στον ε, στόχο του 2010 για τη βιοπικιλότητα ε, και δεσμεύθηκαν μέχρι το 2010 σε μια σημαντική μείωση του τωρινού ποσοστού απώλειας της, της βιοπικιλότητας. Ξέρουμε ότι αυτή η αποτυχία για τη διατήρηση και τη χρήση της βιοπικιλότητας με βιώσιμο τρόπο θα οδηγήσει υποβάθμιση του περιβάλλοντος, νέες ασθένειες, ε, μεγαλύτερη φτώχεια και άνηση ανάπτυξη. Οπότε πρέπει να δράσουμε τώρα για να συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Εμείς ε, στην Επιτροπή μα έχουμε συντάξει προφορική ερώτηση προ το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένα ψήφισμα σχετικά με την διασύνδεση ανάμεσα στην βιοπικιλότητα και την ανάπτυξη εν ώψη τη 11 συνάντηση συνάντησης ε, της διάσκεψης των μερών τη σύμβαση για την Βιοπικιλότητα τη COP10 που θα λάβει χώρα στην ε, στο Αϊτσί της Ιαπωνίας ε, από 18 ως 29 Οκτωβρίου του 2010. Θα εγκριθεί αύριο η προφορική ερώτηση και το ψήφισμα θα υιοθετηθεί στις 5 Οκτωβρίου. υπάρχουν κάποιοι που θα ήθελαν ε, να κάνουν παρατηρήσεις. Μετά θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρίες και κύριοι, γνωρίζω ότι έχουμε χρονικούς περιορισμούς, ότι έχουμε καθυστερήσει σε σχέση με το πρόγραμμά μας. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ, Νέρτζε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ε, καλωσορίζω τη σχέση που αποδίδουμε ανάμεσα στην ε, τη σχέση ανάμεσα στη βιοπικιλότητα, τα οικοσυστήματα και τη σχέση λοιπόν της βιοπικιλότητας με την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Προς το παρόν, και θα περιοριστώ σε αυτό το σχόλιο. Υπάρχουν μόνο δύο αναφορές σε αυτούς τους στόχους της χιλιετίας και θα υποβάλουμε επικοδομητικές τροπολογίες ούτως ώστε να καταδείξουμε με προφανέστερο τρόπο ότι μπορεί να υπάρξουν και αρνητικές όχι μόνο θετικές επιπτώσεις. Αυτά θα ήθελα να πω μόνο. Thank you very much. Ευχαριστώ και εγώ χαιρετίζω αυτή την προφορική ερώτηση και το ψήφισμα διότι νομίζω ότι είναι πολύ καλό ότι η Επιτροπή Ανάπτυξης εξετάζει το θέμα αυτό και θα αντιπροσωπευτεί και στο συνέδριο στην Αγκόγια στην Ιαπωνία. Διότι η αλληλεία είναι ένα από τα μεγάλα οικοσυστήματα τα οποία πρέπει να προωθήσουμε και το ε, η αλληλεία είναι ε, ένα βασικό στοιχείο του εμπορίου από υποανάπτυξη χώρες προς ανεπτυγμένες χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη εισαγωγική αγορά ψαριών και η δεύτερη χώρα είναι η ε, Ιαπωνία που οργανώνει αυτή την ε, αυτό το συνέδριο για τη βιοπικιλότητα. Οπότε θα ήθελα να αφερθώ περισσότερο στους εισαγωγείς αλλιευμάτων, όχι μόνο σχετικά με τη διατροφική ασφάλεια, αλλά και με ε, το υγιές οικοσύστημα και την ε, δυνατότητα ε, τα του θαλασσίου οικοσυστήματος να δεσμεύει το διοξίδιο του άνθρακος που είναι ένα, ε, μία από τις υπηρεσίες που πρέπει να διασφαλιστούν στον κόσμο αυτό. Και υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία θα προσπαθήσουμε να τονίσουμε στις τροπολογίες μας καταρχάς την, αρχή, την αξία του φυσικού κεφαλαίου που δεν εμφανίζεται παρκώς και θα ήταν ε, θανατηφόρο αν οι υποανάπτυξης χώρες δεν μπορούσαν να αναπτυχθούν χωρίς να κάνουν τα ίδια λάθη τα οποία έκανε ο ανεπτυγμένος κόσμος για την εκμετάλλευση και υπερεκμετάλλευση όλων των φυσικών χώρων. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ε, κάποιο τυποποιημένο κριτήριο για να συνδέσει κανείς τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος με οικονομικές αξίες. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να τονίσουμε και στο ψήφισμα αυτό διότι είναι βασικό να προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητα, αλλά είναι κάτι το οποίο τονίζει και την ανεξαρτησία ε, των ε, μικρών ε, παραγωγών και όπως είχε πει πέρυσι ο Όλη που κέρδισε το Νόμπελ της Οικονομίας, ε, είναι βασικό η συλλογική ε, ιδιοκτησία της οικονομίας και των πόρων να ε, εξασφαλίζει και την προστασία της φύσεως και του οικοσυστήματος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άσενς. Αρσένης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι τρόμαξα όταν διάβασα τα πρακτικά της προηγουμένης συζητήσεως για την ε, κατάρτιση της βιοποικιλότητος ε, για την ε, περίοδο μετά το 2020 διότι η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή προσπαθεί να αποδυναμώσει το πρωτόκολλο για την κατανομή των ωφελών. Πρόκειται, φαίνεται να είναι μία νέα πρόταση. Η Επιτροπή λέγει ότι έχει επιφυλάξεις σχετικά με τις γενετικές πηγές και αναφέρεται στις, στους γενετικούς πόρους δεν θέλει να εφαρμόσει το πρωτόκολλο αν ε, δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη και για θέματα τα οποία προηγούνται της υιοθετήσεως του πρωτοκόλου ε, προωθεί την παραδοσιακή γνώση και ούτω καθεξής. Ε, υπάρχει μία συντονισμένη προσπάθεια να αποδυναμωθεί το πρωτόκολλο αυτό, το οποίο ε, είναι απαραίτητο. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι σχετικά με το, με το πρωτόκολλο αυτό στο, σε αυτό το σημείο, διότι θα πρέπει ε, να ε, υπερασπίσουμε και το δικαίωμα όλων των πολιτών ε, να διατηρήσουν τις τοπικές γνώσεις τους. Εγώ θα ήθελα να ακούσω πώς σχολιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα σχόλιά μου. Ευτυχώς, λέει ο Πρόεδρος, δεν υπάρχει κανείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ. Υπάρχει όμως, υπάρχει κάποιος. Α, μάλιστα. Το όνομά μου είναι Γιώργ Ρόρσεν από τη ε, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Δεν εκπροσωπείται η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης δεν μπορώ να σχολιάσω από πλευράς περιβαλλοντολογικής, όχι αναπτυξιακής και να σας πω ότι χαιρετίζουμε το ψήφισμα αυτό. Θεωρούμε ότι είναι κατάλληλη στιγμή να εξετάσουμε το θέμα για να προετοιμάσουμε ε, την συζήτηση για την βιοπικιλότητα που θα έχουμε στη Νέα Υόρκη και νομίζω ότι καλό είναι να συνδυάσει κανείς τα διάφορα θέματα θέματα και θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει και ένα αντίστοιχο ψήφισμα για το COP10 που θα συζητηθεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Προσπαθούμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα που έχουν τεθεί αλλά αυτή τη στιγμή όπου η Επιτροπή είναι εξουσιοδοτημένη για να διαπραγματευτεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα το πράξει. Θα πάω στο τέλος της στο Μόντρεαλ ε, και θα πρέπει να μπορέσουμε ε, να ε, ε, επιφυλαχθούμε ως προς το πώς θα απαντήσουμε όσο δεν έχουμε καταρτήσει την ε, στρατηγική μας και με συγχωρείτε αλλά θα περιμένουμε και θα απαντήσουμε μετά ελπίζω να το αντιλαμβάνεστε τι έχετε να μας πείτε σχετικά με την αποδυνάμωση των πρωτοκόλων Μπορώ να σας πω ότι όπως είπα ε, στις διαπραγματεύσεις αυτές έχουμε ε, τις, ε, τα συμπεράσματα του Μαρτίου 2010 όπου λέγεται ότι υπάρχουν νομικά δεσμευτικά στοιχεία, δεν μπορώ να προχωρήσω περαιτέρω, δεν είμαι ο εμπειρογνώμονος σχετικά με τα πρωτόκολλα αυτά, είναι πράγματα εν τα οποία συζητούνται. Αυτή τη στιγμή αδελφή μου είναι στο Μοντρεάλ και διαπραγματεύονται. Οπότε με συγχωρείτε που δεν μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερες παρατηρήσεις σχετικά με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που επενεύει στο σημείο αυτό, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι και εγώ συμμετέχω στην Επιτροπή Κοινοβούλιο Ευρω... Ε, Ηνωμένα Έθνη και θα ήθελα να έχω τα στοιχεία αυτά διότι ε, διαφορετικά σημαίνει ότι το ένα θεσμικό όργανο θα έχει τα στοιχεία στον ΟΗΕ και το άλλο όχι. Και δεν θα μπορέσουμε να πιέσουμε σωστά για να καταλήξουμε ε, στα σωστά αποτελέσματα σχετικά με τους στόχους της χιλιετηρίας. Θα ήθελα λοιπόν μόλις λάβει τα τελικά πορίσματα η Γενική σας Διεύθυνση να μας τα διαθέσει. Έχουμε ένα πρόβλημα. Ε, η προθεσμία για τις τροπολογίες ήταν την ε, ε, περασμένη Παρασκευή και θα μετατεθεί για αύριο. Αλλά ο κύριος Κάσμαν, ο κύριος Λόβλη θα μπορούσαν να διατυπώσουν ε, τα, τις ε, τροπολογίες στο ψήφισμα που θα συζητηθεί το Σεπτέμβριο στο Στρασβούργο. Αν θέλετε, έχετε ακόμη διαθέσιμο χρόνο. Ωραία. Και τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα. Συνάδελφοι. Α, ήρθαν και καινούργιοι συνάδελφοι. Πολύ ωραία. Τόσο πάντων, περνάει η ώρα και επειδή δεν είναι και πολλοί συνάδελφοι εδώ, Σκέφτηκα να συζητήσουμε τώρα το σημείο 10, την τροπολογία του κανονισμού του Συμβουλίου για σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται για το Γενικό Προπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ω προ την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. You know, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε για τη διαδικασία διαβούλευση για τη συγκρότηση τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο, όπω ξέρετε. Ε, βέβαια, υπάρχουν διάφορα νομοθετήματα που συνδέονται με τη συγκρότηση αυτή τη νέα υπηρεσία και ένα από αυτά συνδέεται και με την τροποποίηση του σχετικού δημοσιονομικού κανονισμού. Οπότε, η Επιτροπή Ανάπτυξη ε, συντάσσει γνωμοδότηση τώρα ε, που θα υποβάλει στην Επιτροπή Προπολογισμών. Ο εισηγητή μα είναι ο κ. Μπέρμαν. Δυστυχώ το κείμενο τη γνωμοδότηση είναι διαθέσιμο στα αγγλικά και μόνο και θα λάβετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τις μεταφράσεις ε, το ταχύτερο δυνατόν. Κύριε Μπέρμαν, θα θέλατε να μας παρουσιάσετε το σημείο. Συγγνώμη, Πρόεδρο. Μιλούσα με τον Ισπανό συνάδελφο. Προσπαθούμε να τα βρούμε με τον Ισπανό συνάδελφο. Είχαμε τον 17ο αιώνα έναν ε, 80 ετών τέλος πάντων πόλεμου. Και στο 117ο λεπτό πήκε το γκολ. Ναι, αλλά έμοιαζε με πόλεμο χθες. As for this. Uh, okay. We are speaking about Μιλάμε για το δημοσιονομικό κανονισμό για την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Αυτή η γνωμοδότηση σχετίζεται με τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα δαπανίσει τα χρήματα και θα ελέγξει τις δαπάνες αυτές. Θα υπάρχει μια σχετική αυτονομία στην ε, διαχείριση του ε, διοικητικού προϋπολογισμού του, της ΕΙΕΒ και το προσωπικό θα έχει διαφορετικό υπόβαθρο της ΑΕΔ και γι' αυτό θα πρέπει εξ αρχής να υπάρχουν πολλές δικλείδες ασφαλείας έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι για την δημοσιονομική ε, ακαιρεότητα. Υπάρχουν, διαφορετικό, υπάρχουν διαφορετικά υπόβαθρα και γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε τις ε, ρήτρες ασφαλείας. Αυτό που προτείνει το αρχικό κείμενο είναι το εξής. Εάν υπάρχει υποψία για οποιαδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο μία καιρότητας θα φτάσει μέχρι την ύπατη εκπρόσωπο. Αλλά θα παραμείνει εκεί. Υπάρχει ε, εσωτερικός έλεγχος, αλλά ίσως το ζήτημα προχωρήσει και περαιτέρω. Θέλουμε να τονίσουμε το ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή και άλλων φορέων που θα μπορούσαν να δουν κατά πόσο υπάρχουν παρατυπίες, όπως η ΟΛΑΦ. Πιστεύω ότι αυτό το κείμενο θα μπορέσει να εγκριθεί χωρίς ε, πολλές ε, τροπολογίες, διότι είναι πολύ απλό και βελτιώνει τη διαφάνεια και την δημοσιονομική ακαιρεότητα εξ αρχής. Και αυτό χρειάζονται οι Ευρωπαίοι πολίτες όταν μιλάμε για δαπάνη των δημοσίων χρημάτων. Θα ήθελε κάποιος άλλος να συνεισφέρει στη συζήτηση. Φαίνεται πως όχι, άρα δίνω το λόγο στην Επιτροπή. Μόλις λάβαμε την έκθεση Μπέρμαν, ο εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμών ε, μόλις ε, έφυγε από την αίθουσα, αλλά επειδή μόλις τώρα λάβαμε την έκθεση μπορούμε να έχουμε λίγο χρόνο πριν επανέλθουμε. Vote on this uh, on, uh, on the 30th of August. Τέλη Αυγούστου είναι η προθεσμία. Okay. Tomorrow morning, uh, immediately στις 10 και 20 μπορείτε να κάνετε την παρουσίασή σας μετά τους συντονιστές δηλαδή και το πρώτο θέμα. Άρα δεν θέλετε να συνοψίσετε, τι να συνοψίσετε. Το επόμενο θέμα είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μπέρμαν για τη θέση του Κοινοβουλίου προς τον προϋπολογισμό του 2011. Αυτή τη βδομάδα το Συμβούλιο θα εγκρίνει τη θέση του για τον προϋπολογισμό του 2011. Έτσι θα ε, εγκριθούν οι τροπολογίες στο κείμενο του Συμβουλίου και έχουμε την δυνατότητα να αποστείλουμε, έχετε δυνατότητα να αποστείλετε ε, τροπολογίες πριν από την 9η ε, Αυγούστου και η ψηφοφορία θα γίνει στις 30 Αυγούστου. Δίνω το λόγο στον κύριο Μπέρμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο προϋπολογισμός του 2011 είναι η πρώτη έξοδος, θα μπορούσαμε να πούμε, της ε, συνθήκης της Λισαβόνας. Ξεκινήσαμε τον Απρίλιο και προβάλαμε τροπολογίες για το τριμερή διάλογο τον Ιούνιο. Ορισμένες από τις ε, τροπολογίες μας ε, λήφθησαν υπόψη ε, ακόμα και σε επίπεδο ολομέλειας. Αυτή τη βδομάδα το Συμβούλιο θα ανακοινώσει τη θέση του για τον προπολογισμό του 2011 και έχουμε ένα προσχέδιο από την Κορεπέρα. Αν λάβουμε υπόψη την χρηματοπιστική κρίση, τε, τις κλιματικές αλλαγές, τους ε, στόχους της ε, χιλιετίας, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι φτωχότερες χώρες δεν θα παραμείνουν εκτός. Ό, να ανακοινωθεί η θέση του Συμβουλίου θα υποβάλω και εγώ τροπολογίες. Θα, η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 9 Αυγούστου και θα ψηφίσουμε στις 30 Αυγούστου. Κλιματικές αλλαγές. Οι κλιματικές αλλαγές δημιουργήθηκαν από τις βιομηχανικές χώρες και δεν θα πρέπει να καταβάλουν το αντίτιμο οι φτωχές χώρες οι αναδύομενες χώρες θα πρέπει να πληρώσουν το αντίτιμο των 100 εκατομμυρίων. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα πακέτο 2,4 δις για τις ε, προσαρμογές στις κρηματικέ αλλαγές. Αλλά τα χρήματα αυτά θα πρέπει να είναι ε, συμπληρωματικά και να μην τα κατακλέψουμε από ήδη υπάρχοντες προϋπολογισμούς. Ως προς το μέσο συνεργασίας αντιτίθεμε να πάρουμε χρήματα από τον τομέα της καταπολέμησης της φτώχειας. Αναφέρομαι στην πρόταση ICI Plus και το DCI θέλει να ελαφρύνει την κατάσταση ως προς τη φτώχεια και όχι να προωθήσουμε τη συνεργασία μας με τις ε, πλούσιες χώρες. Τα 40 εκατομμύρια ευρώ το 2011 που θα βοηθήσουν στους παραγωγούς μπανάνας ίσως ε, προέλθουν από αναπτυξιακούς προϋπολογισμούς μετά από μια συμφωνία στα πλαίσια του ΠΟΕ. Άρα αυτά τα χρήματα θα πρέπει να είναι ε, συμπληρωματικά. Βλέπουμε από την ε, Κορεπέρ ότι ίσως από τον DCI λάβουμε, μάλλον γίνουν περικοπές 16 εκατομμυρίων ευρώ. Ίσως πρέπει να πούμε ότι περικόπτουμε τη γραφειοκρατία, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Επειδή πρόκειται για χρόνια υποτιμημένους τομείς, το Συμβούλιο προβάλλει τη μία πρωτοβουλία μετά την άλλη το Συμβούλιο έχει λιγότερο προσωπικό για να εφαρμόσει το πρόγραμμα ανάπτυξης. Άρα δεν θα πρέπει να γίνουν περικοπές στα διοικητικά έξοδα. Θα πρέπει το προσωπικό να μπορέσει να εφαρμόσει τις πολιτικές που αποφασίστηκαν. Διαφορετικά οι πολιτικές αυτές θα πληγούν ιδιαίτερα. Ε, Επίσης στο Συμβούλιο περιέκοψε 200 εκατομμύρια ευρώ από την επίγουσα βοήθεια. Πρόκειται για χρήματα που χρειάζονται κατεπηγόντως για απρόβλεπτες καταστροφές. Δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε τη στήλη των πληρωμών άδεια, εκτός και αν το Συμβούλιο έχει ειδικέ πληροφορίες και μπορεί να ξέρει ότι δεν θα υπάρχουν κατεπίγουσες περιπτώσεις το 2011. Αυτό είναι ταναστείο, έτσι. Μην το θεωρήσετε κάτι άλλο. Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει την κατάσταση το 2011 και τις ενδεχόμενες φυσικές καταστροφές. Ως προς τη γραμμή για το μέσο δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φαίνεται στις πληρωμές ότι η γραμμή από 90 εκατομμύρια θα μειωθεί σε 60 ε, εκατομμύρια, δηλαδή κατά ένα τρίτο. Είναι πάρα πολλά Ελπίζω ότι η Ευρώπη ε, πρέπει, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο, στην παγκόσμια σκακέρα. Και η Κίνα βεβαίως αλλάζει, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ευθυγραμμιστούμε. Η Ευρώπη βρίσκεται εδώ για να ενισχύσει τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν βλέπω λοιπόν γιατί θα πρέπει να περικόψουμε το εν τρίτον αυτής της γραμμής το 2011. Και θα ήθελα μία εξήγηση από το Συμβούλιο και από την Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε για την πολύ σοβαρή σας εργασία ως προς το, τη σημαντικότερη γνωμοδότηση που έχουμε κάθε χρόνο. Νομίζω ότι και ο συνάδελφος, πρέπει να συγχαρώ και τον συνάδελφο. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να ε, λάβει το λόγο. Διαφορετικά μπορεί να μας ε, απαντήσει η Κομισιόν. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Καλωσορίζουμε πολλά από τα σχόλια που ακούσαμε. Είναι σαφέ ότι πολλές από τις προκλήσεις είναι κοινέ προκλήσεις. Για τις κλιματικές αλλαγές να τονίσω ότι το κονδύλι των 65 εκατομμυρίων για τον προπολογισμό του 2011 προέρχεται ε, απευθεία από τα περιθώρια. Δεν είχε κατανεμηθεί αλλού αυτό το κονδύλιο. Δεν έχουμε πάρει αυτό το κονδύλιο από άλλη γραμμή. Για τα συνοδευτικά μέτρα, για τα 40 εκατομμύρια, ε, λοιπόν, τα 25 τα πήραμε από τα περιθώρια και όχι από άλλες γραμμές. 15 εκατομμύρια ευρώ ανακατανεμήθηκαν ε, και ε, τα πήραμε από άλλα προγράμματα. Δεν έχω τα στοιχεία εδώ ακριβώς από πού προέρχονται, αλλά ανήκουν στην ευρύτερη ανακατανομή των κονδυλίων. Επίσης αναφερθήκατε στη μείωση κατά 16 εκατομμύρια των ε, διοικητικών δαπανών του DCI, του Αναπτυξιακού Οργάνου και όντως ανησυχούμε και εμείς ε, πολύ. 19,4 ε, εκατομμύρια ήταν το συνολικό ποσό και τα 16 τα πήραμε από τα, τις πιστώσεις DCI. Οπότε τα 200 ισοδύναμα σε θέσει απασχόληση όπως ε, ε, ε, τα αποκαλούμε απολέστηκαν και φυσικά μας ανησυχεί πάρα πολύ αυτό. Για την μείωση των πιστώσεων ανάληψη υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν γνωρίζω την κατάσταση που περιγράψατε κανονικά. Αυτές οι πιστώσεις αν, παραδείγματο χάρη, σε επίπεδο ανάληψη υποχρεώσεων είναι στα 19 εκατομμύρια στο σχέδιο προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κανονικά αυτά θα καταβληθούν σε πιστώσει πληρωμών το 2011. Και φυσιολογικά προκύπτουν από υπογεγραμμένε συμφωνίε, οπότε συνιστούν υποχρεώσει. Αλλά θα το εξακριβώσω και θα επανέλθω. Κύριε Μπίρμαν, ε, βρίσκεται ικανοποιητική την απάντηση ναι, το Ευρωπαϊκό Όργανο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα μπορούσατε να το σχολιάσετε επίση για τα 30 εκατομμύρια συμπληρώνει ο πρόεδρο. Ε, ζητώ συγγνώμη. Αυτό εννοούσα στην απάντησή μου. Αν βάλουμε 19 εκατομμύρια ε, στο σχέδιο για τι επιστώσει ανάληψη υποχρεώσεων, αυτό υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι νομικός πώ πρέπει να καταβληθεί σε επιστώσει πληρωμών το 2011. Φυσικά είναι αποτίμηση ε, προς το παρόν. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Εσείς μιλούσατε για μείωση από 30 σε 16 ε, από, αύξηση από 30 σε 60 εκατομμύρια. Πάντω, σε αυτή τη γραμμή του προπολογισμού, ό,τι, ε, υπάρχει σε ανάληψη υποχρεώσεων θα καταβληθεί σε πληρωμή. Πρόεδρος. Για την ε, κρίση για τα τρόφιμα. Έχουμε ήδη ε, κάνει πληρωμές ε, και αναμένεται και άλλη κρίση στην Αφρική. Οπότε ε, τι προβλέπετε να γίνει. Thank you, Mr. Ευχαριστώ. Όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, μείωση είναι που ζητάει το Συμβούλιο. Ξαναλέω, όταν προετοιμάζουμε το σχέδιο προπολογισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε τι τις ανάληψη υποχρεώσεων και αυτό αντιστοιχεί σε ποσά που θα πρέπει νομικώ πώ να καταβληθούν σε σχέση με τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει η Ένωση. Δεν είναι πολιτικό το θέμα. είναι αυτό το ποσό που θεωρούμε εμείς ότι θα πρέπει να καταβληθεί. Αν το Συμβούλιο τώρα έχει αφαιρέσει αυτό το ποσό, δεν ξέρω επί ποια βάσεως έδρασε. Για την έκτακτη βοήθεια, παραδείγματος χάρη, ε, ε, χρειάζεται, να έχουν ε, προβληθεί τα κονδύλια για να γίνουν πληρωμές. Αλλιώς παραβιάζεται τις υποχρεώσεις που έχετε στη συγκεκριμένη σύμβαση. Ε, μιλήσατε για 203 εκατομμύρια, έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω αν το Συμβούλιο πήρε τα λεφτά και τα έβαλε σε αποθεματικό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μάλλον. Θα πρέπει να εξηγήσουν ε, στα λεπτομερή του σχόλιο. Ε, πρόεδρος. Γιατί δεν είναι εδώ το Συμβούλιο. Δεν καταλαβαίνω γιατί σε αυτό το διάλογο δεν είναι όμως ενδιαφερόμενος εδώ. Πρόεδρε, συγγνώμη, ε, το πρόβλημα με τα κατεπήγοντα είναι ότι πρέπει άμεσα να αναλάβετε δράση. Αν δεν υπάρχουν τα κονδύλια, ε, πρέπει να τα βρείτε και χρειάζεται χρόνο. Οπότε Γι' αυτό έχουμε το Ταμείο Έκτακτη Βοήθειας ε, για να έχουμε έτοιμα τα κονδύλια. Δηλαδή το να μα λέτε ότι έχει αναλυθεί υποχρέωση και θα τα βρούμε τα λεφτά. Δεν επαρκεί, δεν είναι αποτελεσματικό αυτό. Είναι μάλλον γελίο. Θα ήθελα το Συμβούλιο να δώσει εξηγήσει. Καταλαβαίνω ότι δεν εκπροσωπείται πάντοτε το Συμβούλιο, αλλά εδώ ε, είναι ενοχλητικό γιατί είναι ε, ε, καθοριστική σε σημασία στο σημείο. Καταλαβαίνω ότι εσείς δεν μπορείτε μάλλον να πείτε κάτι παραπάνω και να μας διαφωτίσετε περισσότερο ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα προσπαθήσω θα προσπαθήσω να ε, μεταδώσω τις απόψεις ε, στο Συμβούλιο, αλλά εγώ συμφωνώ με τις απόψεις σας. Δηλαδή, αν υπάρχει μία γραμμή του προπολογισμού που πρέπει να καλύπτεστε από ε, θα πρέπει ε, να προχωρήσετε γρήγορα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να προχωρήσει πολύ γρήγορα και να σας διαθέσει τα χρήματα. Συμφωνώ λοιπόν με αυτό το οποίο είπατε, αλλά θα προσπαθήσω να δω αν υπάρχει κάποια ενημέρωση από τα έγγραφα που έχουμε από τις τροπολογίες του Συμβουλίου για να προσπαθήσω να καταλάβω γιατί έχει υπάρξει αυτή αλλαγή. Μέχρι εκεί δυστυχώς μπορούμε να πάμε αυτή τη στιγμή, κύριε Μπέρμαν. Κύριε Πρόεδρε, εφόσον μιλάμε για προϋπολογισμό, είναι βασικό θέμα. Το Συμβούλιο θα έπρεπε να εκπροσωπείται. Μπορείτε να στείλετε ένα επίσημο γράμμα διαμαρτυρίας ότι δεν συμφωνείτε καθόλου με την απουσία τους. Ακριβώς αυτό σκόπευα να κάνω και μου είπαν ότι συνήθως το Συμβούλιο δεν, ε, ε, ε, δεν παρίσταται, αλλά εδώ μιλάμε για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο, οπότε γιατί μιλάνε. Θα στείλουμε μια επιστολή στο Συμβούλιο και θα τους πούμε να παρίστανται σε μια... Μου είπαν ότι δεν έχουμε χρόνο τώρα. Κύριε Πρόεδρε, μπορούμε να ζητήσουμε για μια γραπτή απάντηση για την επίγουσα αναπτυξιακή βοήθεια και ε, τα έκτακτα ταμεία. Θα τα σημειώσουμε και ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουν για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε την έκβαση αυτών των θεμάτων τουλάχιστον. Έτσι αντιλαμβάνουμε την κατάσταση, λέει και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Λοιπόν, θα περιμένουμε τότε μέχρι ότου να έχουμε τη γραπτή αντίδρασή τους. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τη γραμματεία επ' αυτού. Νομίζω λοιπόν κύριε Πρόεδρε ότι τελειώσαμε στις 6. Αύριο θα έχουμε τα εξής. Έχουμε σε 9 η ώρα μία συνεδρίαση συντονιστών, μετά θα έχουμε ψηφοφορίες για τις προφορικές ερωτήσεις για τη βιοπικιλότητα στις 10 ε, και στις 10 και 20 θα επανέλθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας μιλήσει ε, για τα οικονομικά εργαλεία που δεν μπορέσαν να παρουσιάσουν σήμερα και στις 11 θα έχουμε μία παρουσίαση της αποστολής στην ΑΕΤ. Σας ευχαριστώ για την, τον τρόπο με τον οποίο μας παρακολουθήσατε. Η συνεδρίαση διακόπτεται. Ευχαριστώ.